Now let's go. Λοιπόν, έδωσα άλλα δύο λεπτά. Ελπίζω να απολαύσατε το γεύμα. Work Και ίσως και άλλες εργασίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατάφερα να έχω πέντε συναντήσεις. Remarkable. Αξιοσημείωτο τι μπορεί να κάνει κανεί όταν εργάζεται. Κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Επιστρέψαμε. Να σας πω τι έγινε συνεδρίες των συντονιστών. Δεν έχουμε πολλά μέλη παρόντα. δεν είναι εδώ θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Εγκρίναμε το σχέδιο μερίσας διάταξης για την 28 Ιανουαρίου. Αυτό είναι το πρώτο. Και εγώ θα είμαι συγκήτρια για γνωμοδότηση για την εφαρμογή, της, για την εφαρμογή ε, του κοινοτικού δικαίου, ετήσια έκθεση 2014, σύμφωνα με το σύστημα DEONT. Αλλά ανταυτού θα διοριστεί υποψήφιο την για την ευρωπαϊκή προσβασιμότητα εξαιρετική πράξη, κατόπιν αιτήματο των πολιτικών ομάδων, συμφωνήσαμε με κατόπιν αιτήματο των Πρασίνων να αφήσουμε την αναφορά 1771 του 2013 ανοιχτή και να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίε από τι Ισπανικέ Αρχέ. Επίση, οι συντονιστέ συμφώνησαν με το αίτημα του ΕΛΚ να αποσυρθεί μια αναφορά η 1270 του 2014 ένα αίτημα του ΕΛΚ να κλείσει, να 43 αναφορές αμφισβητήθηκε από άλλες ε, ομάδες και συμφωνήθηκε ότι η Γραμματεία θα κάνει την αξιολόγηση των αναφορών και θα τη συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη τις επόμενες μέρες οπότε αυτό είναι δυνατόν. Κατόπιν αιτήματο του EFTD να εφαρμοστεί τη δικασία κατεπηγόντως στις αναφορές τυπου οι συντονιστές συμφώνησαν ότι η κανονική διαδικασία περί αναφορών θα ισχύσει και η γραμματεία θα ομαδοποιήσει τις αναφορές του TTIP μαζί ούτως ώστε να μπορούσαν να ενταχθούν σε μελλοντική ατζέντα σύντομα λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από μερικούς μήνες ε, είχαμε μία γνωμοδότηση επί του θέματος οπότε αυτό λοιπόν εντάσσεται στην κανονική διαδικασία για, για, για συστάσεις εγκρίθηκαν οι συστάσεις μου ε, όλες εκτός από τρεις ε, περιπτώσεις οι οποίες θα κοινοποιηθούν στα πρακτικά αναφορά 0177 του 2015 αναφορά 0199 του 2015 και 0214 του 2015 όσον αφορά τις επισκέψεις ε, στην Ισπανία από 8 με 10 Φεβρουαρίου έξι μέλη και τρία μέλη εξ ανακοίνωσαν ότι θέλουν να μπουν στην αποστολή και έχουν δεσμευτεί να υπάγουν. Ε, οπότε αυτό θα πρέπει πραγματικά να υπογραμμιστεί. Οι συντονιστέ συμφώνησαν ότι ο αντιπρόεδρος ε, της, ε, του ΕΛΚ, θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας και αποφασίσαμε στη δημόσια ακρόαση και ζήτησα από τους συντονιστές όσον αφορά το θέμα να προτείνουν ονόματα για ομιλητές που θα συμμετάσχουν στην ακρόαση και αποφάσει επί των ονομάτων και του προγράμματος θα ληφθούν μέσω γραπτής διαδικασία, αρχές Ιανουαρίου. Φαίνεται κάτι απόμακρο, αλλά λίγες εβδομάδες μας χωρίζουν τις αρχές Ιανουαρίου. Όσον αφορά τι προφορικέ ερωτήσει, την προφορική ερωτήση για τη συνθήκη του Μαρακέ, οι συντονιστέ συμφώνησαν να υποβάλουν σύντομο ψήφισμα τη Επιτροπή Αναφορών στην Ολομέλεια επ' αυτού να εφητηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής τον Ιανουάριο και τα άλλα σημεία 8, 9, 10, 11 και 12. Έχετε τις πληροφορίες στους φακέλους σας για τα διάφορα συντονιστές ε, λένε ότι θα παραχθεί ένα, ένα, θα ένας φάκελος με έντυπα από τον Ιανουάριο κατόπιν ετήματο, διότι θέλουμε τελικά να μην χρησιμοποιούμε πια χαρτιά στις εργασίες τη Επιτροπής αυτό συμφωνεί με το αίτημα και τη πάρα πολλών πολιτών επιθυμία και να φύγουμε από τον αναλογικό κόσμο και να επιλέξουμε τον ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας και έτσι εργαζόμαστε και εκείνους σαν και εμένα που είναι κάπως διστακτικοί σίγουρα θα μας δοθούν οι αναγκαίες πληροφορίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει χωρίς έγγραφα χαρτιά. Λοιπόν πρέπει μέχρι 19 Ιανουαρίου να ζητήσετε αν θέλετε χαρτιά, τα έγγραφα σε χαρτιά και αυτό θα ισχύει για το επόμενο έτος. Να λαμβάνετε τα έγγραφα σε χαρτί, αν το ζητήσετε και υποσχέθηκε η γραμματεία να μας το υπενθυμίσει όταν θα επιστρέψουμε μετά τις γενιάτικες διακοπές. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ε, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να κινηθούμε και να πάμε στην πρώτη αναφορά του Κωνσταντίνου Γιανόπουλου όσον αφορά θέμα κυδαιμονίας παιδιού. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που παρίσταστε. Γνωρίζουμε την υπόθεση και θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε, έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη με το απόγευμα. Καταρχάς το λόγο δίνουμε στον αναφέροντα για πέντε λεπτά και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στα μέλη. Παρακαλώ όσο μπορείτε να είστε σύντομος αν έχετε την καλοσύνη. Και έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Αφορά την απαγωγή παιδιού, αν μπορώ να το διορθώσω. Δεν αφορά θέμα επιμέλειας παιδιού. Την, την Λοιπόν, αν αναφερόμαστε στον πώ μπορούν να εκδίδονται διαβατήρια χωρί την ε, συνένεση των γονέων. Εκεί έχουμε παραβίαση της Συμφωνίας Βρυξελών 2 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι η έκδοση του διαβατηρίου δεν εμπίπτει στο πεδίο του κανονισμού. στι 21 Οκτωβρίου του 2015 ε, εξεδόθη απόφαση του δικαστηρίου υπαριθμών C215 του 2015 που λέει ότι η έκδοση διαβατηρίου για ανηλίκους εμπίπτει στο υλικό πεδίο του κανονισμού Βρυξέλλες 2 και απαιτείται συνένεση όλων εκείνων που έχουν γονική ευθύνη. Ε, είναι σαφές λοιπόν, υπήρχε αυτός ο κανόνας, αυτή η απόφαση από το 2005 όταν ετέθησε ισχύ, ε, σε ισχύ η Βρυξέλλες 2. Τρεις μέρες αργότερα ήρθα σε επαφή με το, γραφείο Εκτό διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και είπαν ότι εμένα στην απόφαση του 2015 που ανανέωσαν τα διαβατήρια και θα πρέπει να φέρουν απόφαση του δικαστηρίου για να σταματήσει η έκδοση διαβατηρίου. Πρέπει να δουν την έκδοση του διαβατηρίου, την απόφαση του δικαστηρίου για να μην εκδώσουν διαβατήριο χωρίς τη συνένεσή μου και αυτό δεν είναι δυνατόν. Πέραν αυτού θα ήθελα να επενθυμίσω στο Κοινοβούλιο και το εξής ότι ο κανονισμός 444 2009 που αφορά το Σέγγεν, το κανονισμούς Σέγγεν, άρθρο 1, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια έκθεση περί εναρμονίσεως των κανόνων για παιδιά που ταξιδεύουν έξω από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών και για την ασφάλεια αυτών. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη το Κοινοβούλιο να εναρμονίσει τους κανόνες. Το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι κανένα παιδί, κανείς κάτω των 18 δεν μπορεί να λάβει το δικό του διαβατήριο χωρίς τη συνένεση όλων εκείνων που υπέχουν γονική ευθύνη. Πιθανότατα αυτό θα επέλυε το πρόβλημα όλων των παιδιών που πηγαίνουν να πολεμήσουν στη Συρία και που πεθαίνουν εκεί χωρίς τη συνένεση όλων εκείνων που υπέχουν γονική ευθύνη η έκδοση των διαβατηρίων των δύο παιδιών το 2010 βοήθησε ε, τη μητέρα να τα πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα πάρει σε τρίτη χώρα. Ήταν διοικητική η απόφαση των Εθνικών Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου που παραβιάζουν τα όρια του κράτους δικαίου και είναι συνεπώς παράνομη απόφαση. Οπότε τα διαβατήρια των παιδιών μου είναι αυθεντικά αλλά παράνομα. τα κεκτημένα Σέγγεν και Βρυξέλλες διετονίζουν τονίζουν ότι εκείνοι που ταξιδεύουμε νόμιμα πρέπει να ταξιδεύουμε νόμιμα εξωτικά έγγραφα μεταξύ κρατών μελών. Οπότε επαφίεται, στην απόφαση του Κοινοβουλίου επ' αυτού. Υπάρχουν κάποια επίμαχα ζητήματα ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει ότι ο κανονισμός δεν καλύπτει τις, τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να εκδοθεί παιδικό διαβατήριο, διότι αυτό είναι θέμα που αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Είναι λανθασμένη αυτή η δήλωση που έγινε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πολίτες της Ευρώπης. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σίγουρη πώς ε, να ερμηνεύσει τον νόμο, μπορεί να έχει επιφυλάξει να παραπέμψει το θέμα στο δικαστήριο. Όχι να προβαίνει σε τις δηλώσεις όπως αυτές που μόλις προανέφερα τώρα. Αυτό θέτει ένα θέμα. Μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ε, εκθέσεις που αφορούν αναφορές ε, πολιτών. Όσον αφορά την απαγωγή στην Κύπρο, θα θυμόσαστε στην προηγούμενη ακρόαση ότι υποφασίστηκε ότι η Επιτροπή θα στείλει ε, επιστολέ στο Υπουργείο μαζί με εξώδικα έγγραφα, το εξώδικο έγγραφο που είχα προσαρτήσει στην αναφορά μου και να ζητήσει απαντήσεις για κάποιες ερωτήσεις. Ο Υπουργός απάντησε μετά από ένα εξάμεινο και μετά από κάποια τηλεφωνήματα από τη Γραμματεία και βασικά είπε ότι η υπηρεσία του έχει εκτελεστική εξουσία και μόνο και απόφαση να μην συνεχιστούν οι κλιματικές έρευνες στην απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα που αποτελεί ξεχωριστό φορέα, ανεξάρτητο φορέα. Πρέπει να πω ότι ο Ισαγγελέας δεν εκπροσωπείται διεθνώς ο ίδιος αλλά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ίσως ο ανεξάρτητος φορέας, ο Ισαγγελέας είναι ανεξάρτητος φορέας στη χώρα αλλά δεν εξωγενής όσον αφορά το κάτω δικαίου και δεν είναι υπέρτερος του κράτους δικαίου και πρέπει να απαντήσει ε, στις ερωτήσεις που τα απευθύνονται. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή να στείλει εκ νέου την επιστολή αν θέλει αμέσως, άμεσα στον Ισαγγελέα και να ζητήσει να απαντήσει στο εξώδικο έγγραφο αυτό που έλαβε το Δεκέμβριο του 2013 του επεδόθη νομίμως και ακόμα αναμένεται απάντηση. Θα ήθελα να ζητήσω να επεκταθεί η έρευνα και να καλύψει και την Ελλάδα. Το ζήτησα αυτό, αλλά στη δίκη πριν πάνω ένα χρόνο για τη δίκη του διαζύγιο στην Αθήνα ετέθη θέμα δικαιοδοσίας και μας ζητήθηκε να, να θέσουμε ε, στο δικαστήριο ε, μία ερώτηση για ε, προδικαστική απάντηση. Τώρα, τώρα είναι και το θέμα της δικαιοδοσίας. Ο κανονισμός αναφέρεται στις εθνικούς κανόνες και μόνο πρέπει την κατάλληλη στιγμή να εφαρμόζεται εθνικοί κανόνες και δεν εφαρμόζεται εθνικοί κανόνες ανεξάρτητα αλλά σαν κανόνες εντός του πλαισίου του κανονισμού. Υπήρξε κάποια πολιτική παρέμβαση εκεί και η απόφαση μετά από 15 μήνες εκρεμεί ακόμα και δεν παρεπέμφθη στο ΔΕΚ το θέμα. Λοιπόν, για τη σωστή απόδοση δικαιοσύνης, είτε να εκδοθεί απόφαση, ας αποσταλεί το θέμα στο ΔΕΚ, διότι έχει παράλληλες συνέπειες για το θέμα της ε, επιμέλειας των παιδιών. Μπορεί να εκκρεμεί επί 10 χρόνια ή περισσότερο. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε μια απόφαση και στις δύο υποθέσεις. Δεν μπορεί να καθυστερεί η απόφαση, διότι ένας πολιτικός κάποιο υπουργό δεν του αρέσει το θέμα αυτό και δεν του αρέσει η ερώτηση. Και είμαι σίγουρο ότι πολλοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι την ερώτηση, η οποία όμω πρέπει να απαντηθεί. Λοιπόν, ποια είναι η παρούσα κατάσταση. Το θέμα είναι στο Eurojust. Τα παιδιά έφυγαν ε, το καλοκαίρι, έλειπαν, τους βάλαμε στο σύστημα SIS, τους ψάξαμε, υπάρχουν λεπτομέρειες έχουν εντοπιστεί ότι είναι στην Ουγγαρία, του συνετόπισε η αστυνομία, ταξίδεψα, τα συνάντησα τα παιδιά, δεν μπορούν να βγουν από το χώρο Σέγγεν. Επί προσωρινής βάσης έμεναν εκεί, εξέπνευσε η παραμονή, έμειναν πάνω από τριμηνού. με διαβατήρια που δεν έχουν εκδοθεί νομίμως όπως σας είπα, παρεπάμψαμε το θέμα στο Eurojust. Θα ήθελα το Eurojust να συντονιστεί με τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται και αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κρατών μελών ε, υπάρχουν νομικές υπηρεσίες που μπορούν να τοποθετηθούν. Θα ήθελα λοιπόν το Κοινοβούλιο να στείλει επιστολή στο Eurojust ζητώντας το Eurojust να εξετάσει με ανοιχτό τρόπο την υπόθεση και να αποφασίσει σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Τέλος, πέρσι απεστάλλει επιστολή προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να φτάσουν στην πρεσβεία και να έχουμε απάντηση. Τον περασμένο Οκτώβριο είχαμε κάποια απάντηση. Θέλω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η δυνατότητα, ο διπλωματικό διάλογο, διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η μητέρα να επιστρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, διότι δεν έχει δουλειά στην Ουγγαρία που, ε, που ζει και εξαρτάται από την επιχείρησή της την οποία την διευθύνουν άλλα μέρη ε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, θέλω να παραμείνουν όλοι, όλες οι διέξοδοι ανοιχτέ, ούτω ώστε να βρεθεί μια διπλωματική, μια λύση τελικά στο όλο θέμα. Να μείνουν όλα ανοιχτά. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο Και τώρα α δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή, τον κύριο Γκρούμπισιτ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα ε, που μας ανέφερε όλα αυτά τα θέματα για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε σήμερα και ελπίζω να τα διευκρινίσουμε. Πρώτον, όπως τόνισε ο αναφέρον, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C215 του 2015 ε, που αφορά τη συνένεση των γονέων για να εκδοθεί διαβατήριο για ανήλικο παιδί. Ε, είμαι υποχρεωμένος να διαφωνήσω με τον αναφέροντα. Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αυτή η απόφαση δεν σημαίνει, δεν ορίζει ότι θα πρέπει να είναι παρόντες και οι δύο ε, γονείς ή να έχουν χορηγήσει ε, ρητά τη συνένεσή τους και την άδειά τους. Για να το διευκρινίσουμε, ελπίζω να με να μπω λίγο στο κείμενο της απόφασης, για το σημείο 15, στην παράγραφο 15 της απόφασης, ε, ορίζει το δικαστήριο σαφώς ότι με βάση το βουλγαρικό νόμο οι αποφάσεις για τα διαβατήρια θα πρέπει να λαμβάνονται με κοινή συνένεση των γονέων και συμφωνία. Είναι γεγονός ότι αναφέρει ένα στοιχείο ότι θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν δώσει την άδειά τους, ε, αλλά αυτό αναφέρεται στο βουλγαρικό δίκαιο. Αυτό το προπετούμενο είναι του βουλγαρικού νόμου, να έχουμε την άδεια και των δύο γονέων. Όπως είπε και ο ίδιος ο αναφέρον ε, πριν από λίγο, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου είπαν ότι η εθνική τους νομοθεσία ορίζει ότι αρκεί ένας μόνο γονέας να το ζητήσει και εκδίδεται το διαβατήριο. Ε, η απόφαση την οποία επικαλείται και παραθέτει ο, ο αναφέρον μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν το προβλέπει, το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, δηλαδή ότι χρειάζεται να ε, συμφωνήσουν και οι δύο γονείς. Τότε και μόνο τότε μπορεί να ισχύσει αλλά όχι ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η θέση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια είναι ότι η απόφαση αυτή και η νομολογία που παρουσιάζει ο αναφέρον δεν έχει σχέση με την περίπτωση αυτή και παραμένει στην άποψή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την Κυπριακή νομοθεσία και τη διαδικασία ε, που κρεμεί στην ελληνική δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μελετήσει αυτά τα θέματα και έχει καταλήξει σε μία γνώμη και παραμένουμε σε αυτή τη γνωμοδότησή μας που λέγει ότι εδώ δεν εφαρμόζεται καμία κοινοτική ευρωπαϊκή νομοθεσία από την έννοια που ε, επικαλείται ο αναφέρον και δεν μπορεί να επέμβει σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. I thank you very much and I'm... Σας ευχαριστώ πολύ να καλέσω τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην ε, συζήτηση. Ελεονόρα Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προφανώς χρειάζεται και άλλο επίπεδο ερμηνεία. Και εγώ έχω εδώ μπροστά μου την απόφαση του δικαστηρίου. Στο τελικό κομμάτι, στο τελικό τμήμα δηλώνει το δικαστήριο. Αν μπορώ να διαβάσω. Η δράση με την οποία ένας από τους γονείς ζητά από το δικαστή να καλύψει την έλλειψη συνένεσης ε, του άλλου γονέα για τη μετακίνηση των ανηλίκων. Παρακαλώ, Ελεονόρα, μπορείς να ξαναρχίσεις, διότι δεν ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπες. Πιο σιγά. Να έχουν και κάποια τύχη διερμηνής. Εν πάση περιπτώσει, στο τελικό τμήμα της απόφασης το δικαστήριο δηλώνει ότι η δράση με την οποία ένας από τους γονείς ζητά από τον δικαστή να ξεπεράσει την έλλειψη συνένεση του άλλου γονέα όσον αφορά τη μετακίνηση των ανηλίκων εκτός του κράτους μέλους διαμονής του ιδίου και την εκχώρηση έκδοση ενός διαβατηρίου στο όνομα αυτού εμπίπτει στην ε, σφαίρα ε, ε, του 22.0 του κανονισμού 22.01 του 2003 δηλαδή Βρυξέλλες 2 Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ συχνά χανόμαστε στις ερμηνείες και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μία απάντηση ενδελεχέστερη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που κατά την άποψή μου ε, που δεν η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν ικανοποιητική. Θα ήθελα να στραφώ και προς τη φράση που ο αναφέρον χρησιμοποίησε πριν στις διαφάνειες που έδειξε. Τα παιδιά του έχουν διαβατήρια αυθεντικά αλλά παράνομα είπε. Κατά την άποψή μου είναι με εμφράση που συνοψίζει άριστα τις συνθήκες υπό τις οποίες πάρα πολλές οικογένειες βρίσκονται και ζουν τέτοιες συνθήκες, τέτοιες καταστάσεις αβεβαιότητας και αντίφασης, ακραίες αντιφέστασης μέσα στα πλαίσια των κενών της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Χάνονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει να αποσαφινιστεί το όλο θέμα και μία από τις δράσεις που αναφέρον πρότεινε, δηλαδή να, να αποσταλεί μία επιστολή και να ζητηθεί από την Κύπρο μία απάντηση σαφής, ακριβής, χωρίς να κρύβονται πίσω από τυπικές διαδικασίες, χωρίς να επομίζονται τις ευθύνες των δράσεών τους, να γίνει, να αποσταλεί αυτή η, επιστολή από την Επιτροπή Αναφορών, να ζητηθεί δηλαδή μια απάντηση από τις Κυπριακές Αρχές. Ούτως ώστε να δοθεί συνέχεια σε αυτή την υπόθεση που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Και τέλος, και η έκκληση των αφέροντος να ανοίξουν και διπλωματικές επαφές με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι κάτι που σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει, πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Και από την Επιτροπή Αναφορών εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε το αίτημα του αναφέροντος γι' αυτό. Κατά την άποψή μου αυτή είναι μια αναφορά που θα πρέπει να παραμείνει προφανώς ανοιχτή διότι καλύπτει πολυάριθμα προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα που βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Βλέπουμε και το πώς υπάρχουν οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες και πώς εφαρμόζεται αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία στα κράτη-μέλη και υπάρχουν προβλήματα από την υλοποίηση του κοινοτικού δικαίου στα κράτη-μέλη. Κυρία Ντανόκα, παρακαλώ. κυρία Ντανόκα. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα γιατί επιμένει ε, στην υπόθεσή του γιατί μέσω αυτών των πολύ συγκεκριμένων υποθέσεων ε, εμεί ε, ω συνομοθέτες και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να καταλάβουμε πού υπάρχουν κενά στην νομοθεσία μας και ειδικότερα στον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Γνωρίζουμε ότι Είμαστε σε θέση τώρα ε, να επηρεάσουμε τη διαδικασία τροποποίησης ε, του Βρυξέλλες 2 και θα λάβουμε υπόψη το πρόβλημα που παρουσιάζεται και στη δική σας ε, υπόθεση και που έχει να κάνει επίσης ε, και με την έλλειψη ε, της, ε, της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Πέρσι ήταν το ευρωπαϊκό έτος της ηθαγένειας και είχαμε μάλιστα και ολόκληρη έκθεση στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Όμως δυστυχώς Όταν ε, μιλούμε για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, το μόνο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται είναι η άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αλλά δεν μιλούμε για το πρόβλημα για, την, για το γεγονός ότι ε, η ευρωπαϊκή ηθαγένεια μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία ε, σε σχέση με την ηθαγένεια κάποιας χώρας. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων νομοθεσιών. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία χρειάζονται, χρειάζεται συμφωνία και των δύο γονέων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται συμφωνία του ενό μόνο. Χρειάζεται μόνο ένα γονέα. Δεν ξέρω ακριβώ τι γίνεται στην Κύπρο. Υποθέτω ότι στην... στην Κύπρο και οι δύο γονεί πάλι χρειάζονται. Μάλιστα. Σε αυτέ λοιπόν τις δασυνοριακέ υποθέσεις πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση τη νομοθεσία όσον αφορά την ηθαγένεια των παιδιών και αν γινόταν αυτό νομίζω θα ήταν καλό και ίσως προς αυτήν την ε, κατεύθυνση θα μπορούσαμε να κινηθούμε όσον αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κοιτάξτε, και εγώ Ήμουν ε, εισηγήτρια για μία ε, έκθεση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία για να υπάρξει ελεύθερο καθεστώς χορήγησης ε, θεωρήσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ώστε να υπάρξει ενδεχομένως καλύτερη συνεργασία με τη χώρα αυτή. Ίσως και εδώ να φαίνεται ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας με τη χώρα αυτή. Ε, καταλαβαίνω επίσης και την επιχειρηματολογία της κυρίας Εύη ότι δεν είναι διεξοδική η επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό θα ήθελα να διατηρηθεί ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά για να γίνει καλύτερη αξιολόγηση της υπόθεσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ο αναφέρον νομίζω ότι εκτεταμένα παρουσίασε την υπόθεσή του και θα έλεγα και το προσωπικό του δράμα, διότι είναι δεδομένο ότι έχει στερηθεί τα παιδιά του. Και αυτό βεβαίως ε, είναι ένα θέμα ηθικό, συναισθηματικό, αλλά άπτεται και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα γιατί ο αναφέρον είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερο θα έλεγα ότι εμείς πρέπει να δούμε και από μια άλλη σκοπιά το, το συμφέρον των παιδιών και ιδίως του ανήλικου παιδιού διότι ε, ταυτόχρονα έχει την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Επομένω επανέρχομαι σε αυτό που είχα πει και άλλη φορά ότι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια αποτελεί τον πυρήνα, τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε για να δούμε ορισμένα θέματα οικογενειακού δικαίου διότι το οικογενειακό δίκαιο δεν εμπίπτει ως τέτοιο στενά στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ξεκάθαρα μια αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως, από τη στιγμή που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, θα πρέπει να δούμε μήπως πλευρές του αστικού δικαίου, του οικογενειακού δικαίου, επηρεάζουν τα δικαιώματα όσων έχουν ευρωπαϊκή ηθαγένεια, άρα είτε των γονέων είτε των παιδιών και επομένως εγώ θεωρώ ότι εκεί είναι η καρδιά όλου του θέματος που μπορεί να μας βοηθήσει και στην υπόθεση αυτή και σε άλλες υποθέσεις που εξετάζουμε. Δεν ε, κρίνω ε, ικανοποιητική την απάντηση της ε, Επιτροπής και νομίζω ότι αυτό εκτέθηκε και από τις συναδέλφους. Υπάρχουν τρία-τέσσερα σημεία που μπορούμε να θίξουμε. Πρώτον, είναι δεδομένο ότι έχει εμπλακεί η Eurojust και επομένω, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Εμείς ως Επιτροπή θα μπορούσαμε να κρατήσουμε πρώτα απ' όλα την υπόθεση αυτή ανοιχτή, να ζητήσουμε επιπλέον πληροφόρηση από την Eurojust και την παρέμβασή της σε ένα θέμα καταγγελίας που έχει γίνει και έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες νόμιμα μέσω των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών για να φτάσει το θέμα στη Eurojust. Άρα λοιπόν ένα θέμα το οποίο βάζουμε μπροστά. Δεύτερο θέμα. Υπάρχει ένα ζήτημα που νομίζω θα μπορούσαμε να απευθύνουμε επιστολή στη μόνιμη αντιπροσωπεία τη Ουγγαρία. Γιατί υπάρχουν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με το τι θα γίνει με την εξέλιξη αυτών των παιδιών, αν θα πάρουν άδεια παραμονή, αν μπορούν να πάρουν άδεια παραμονή, τα θέματα που έθεσε ο αναφέρον, η εμπλοκή της Eurojust. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρο ένα θέμα που αφορά την Ουγγαρία και νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθεί και να έχουμε και την άποψη της Ουγγαρίας. Το τρίτο θέμα είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε μια καλύτερη απάντηση και από τις Κυπριακές Αρχές. Καταλαβαίνω ότι οι Κυπριακές Αρχές θεωρούν το ζήτημα ξεκάθαρο μιας δικαστικής δικαιοδοσίας, επομένως σου λέει ότι ως κράτος δεν μπορώ να παρεύω, όμως νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια επαφή και με την Κυπριακή πλευρά για να δούμε πώς εξελίσσεται η υπόθεση. Το τέταρτο, είμαι σύμφωνος ότι δεν μπορεί στα Αραβικά Εμμυράτα ή σε όλες αυτές τις αραβικές χώρες να υπάρχει μια κατάσταση γκρίζας ζώνης, όπου πάνε και κάποιοι δεν εφαρμόζονται νόμοι και χάνονται τα ίχνη. Λοιπόν, να υπάρχει η δυνατότητα και νομίζω κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε θα μπορούσαμε να απευθύνουμε μία νομιζω κυριε κυρια προεδρε θα μπορουσαμε να απευθυνουμε μια επιστολη και στα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα λοιπόν κλείνοντας θεωρώ ότι η υπόθεση πρέπει να μείνει ανοιχτή ως αναφορά, να κάνουμε αυτές τις επιστολές και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε μια υπόθεση όχι υπέρ του συμφέροντος, θα έλεγα του αναφέροντος ή της συζύγου του, αλλά να δούμε το συμφέρον των παιδιών. Διότι έχουμε μια μονομερή αυτή τη στιγμή δραστηριότητα του ενός γονέως, όπως εκτιμά ο γονέας αυτός ή η σύζυγος την έννοια του συμφέροντος των παιδιών, αλλά αυτό είναι κάτι υποκειμενικό. Εμείς πρέπει να δούμε το αντικειμενικό θέμα. Ε, επομένως θεωρώ ότι παρότι έχει πολλές νομικές πλευρές οι οποίες ε, πρέπει να εξεταστούν και δεν είναι εύκολο να εξεταστούν όμως από πλευράς δικής μας μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πέντε βήματα τα οποία βλέπω συμφωνούν και οι συνάδελφοι ήδη τα είπαν πριν ούτω ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε για να έχουμε μια ε, ευνοϊκή εξέλιξη της υπόθεσης αυτή. αυτής. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ντάλινγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να καθυστερήσω τη συζήτηση περισσότερο από ό,τι πρέπει. Απλώς να πω ότι μερικές φορές ε, σε έτσι πολύ κρύα και καθαρά ε, νομικά υπάρχει μία ε, αλήθεια σε όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρέθεσε μία πολύ λεπτομερή αιτιολόγηση για, το πώς, για, τα, για τους περιορισμούς της νομοθεσίας. Από την άλλη όμως υπάρχει και η πραγματικότητα της κυκλοφορίας των ανθρώπων και ε, το, οι διεθνείς και η πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων δεν συνάδει με αυτήν την ε, ε κρύα ανάγνωση ε, της νομοθεσίας. Έτσι είναι τα πράγματα και αυτή είναι η πραγματικότητα με την νομοθεσία. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε η Ελεονόρα Εύη. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει αυτή η αναφορά ανοιχτή. Πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες και θα έπρεπε επίσης ε, να ε, γράψουμε, να αποστείλουμε μία επιστολή στις κυβερνήσεις ε, τις οποίες αφορά αυτή η υπόθεση. Ίσως να τις συμπεριλάβουμε αυτές τις συζητήσεις και στην ομάδα εργασίας για την ευημερία των παιδιών, επειδή θα υπάρξει και μία προφορική ερώτηση γύρω από τον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Αυτό θα προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο στη συζήτηση αυτή όσον αφορά την προστασία των παιδιών και τις Βρυξέλλες 2. Θα ήταν νομίζω σφάλμα να κλείσουμε την αναφορά αυτή πριν γίνει αυτή η συζήτηση ε, στην Ολομέλεια γύρω από τον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ πολύ είναι μια υπόθεση που πολλές φορές έχει εξεταστεί και λόγω της παρούσας νομοθετικής κατάστασης δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Οι εργασίες για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 εκκρεμούν. Δύο ζητήματα υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα η έκδοση εγγράφων. Αυτό είναι τμήμα των εθνικών αρμοδιοτήτων και Αμφιβάλλω κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν ποτέ ότι τέτοιου είδους έγγραφα πρέπει να εκδίδονται επί τη βάση διεθνών διατάξεων. Αλλά όσον αφορά την ε, συνένεση των γονιών για το ταξίδι των παιδιών σε μερικές ε, χώρες ε, χρειάζεται η, συνένωση, η συνένεση και των δύο γονέων και σε άλλες χώρες χρειάζεται απλώς ένας γονιός να αποφασίσει. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία. Ε, ίσως είναι τμήμα της κουλτούρας της κάθε χώρας. Στις χώρες στις οποίες ε, χρειάζεται συνένεση των δύο γονέων, συμβαίνει ένας γονέας να μπλοκάρει, να παρεμποδίζει την απόφαση και ενδεχομένως να είναι αδύνατον για τα παιδιά να εγκαταλείψουν ε, τη χώρα. Γιατί ένας γονιός με το παιδί του δεν μπορεί ας πούμε να προχωρήσει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία επειδή κάποιος άλλος γονιός δεν του επιτρέπει να ταξιδέψει με τα παιδιά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι μπορούμε να επιτύχουμε αφήνοντας αυτήν την αναφορά ανοιχτή. Εγώ νομίζω ότι απλώς θα είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας οι πολιτικοί πρέπει να δώσουν ελπίδα στον κόσμο ότι μπορούν να τους βοηθήσουν, αλλά βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Οπότε ας είμαστε, ας είμαστε ειλικρινείς. Μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε σε αυτή την περίπτωση με την ε, υφιστάμενη νομική κατάσταση. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, αν μου επιτρέπετε θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ζήτημα. Βεβαίως η εναρμόνιση, όπως είπε η κυρία Σδάνοκα, ε, είναι πραγματικά στο ευχολόγιο κάθε Ευρωπαίου φεντεραλιστή. Δυστυχώς όμως απέχουμε πόρο από αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς κατ' σύμφωνα με τη δική μου άποψη και το διευκρινίζω. Ε, η έκδοση διαβατηρίων ε, είναι στην επικουρικότητα. Με άλλα λόγια, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα παρά να ε, αγωνιστούμε για να έχουμε περισσότερο φεντεραλισμό στην Ευρώπη και σε αυτά τα θέματα. Βέβαια αυτό δεν σας βοηθάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, ούτε τον αναφέροντα, ούτε τα παιδιά. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, γιατί θα σας δώσουμε το λόγο σε λίγο, να μας πείτε, να σας ρωτήσω, υπήρξαν κάποιες εξώδικες ε, απόπειρες να λυθεί το πρόβλημα σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει δυνατότητα διαμεσολάβησης μεταξύ των δύο γονέων που δεν ε, μιλάνε ο ένας τον άλλον, που δεν συνεννοούνται και δεν επικοινωνούν και δεν συμφωνούν για την επιμέλεια των παιδιών τους και τη γονική μέρη. Υπήρξαν απόπειρες τέτοιες συμφιλίωσης μεταξύ των δύο γονέων και διαμεσολάβησης και επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Μαριάς, διότι αυτό που έχει πραγματικά σημασία και είναι ο πυρήνας αυτής της Επιτροπής είναι το συμφέρον των παιδιών το καλύτερο για τα παιδιά. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το καλύτερο ε, συμφέρον, το καλό ενόμενο συμφέρον των παιδιών είναι να έχουν καλή σχέση και με τους δύο γονείς, όταν ζουν και οι δύο γονείς. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις τραγικά ε, έχουν ένα γονέα μόνο, τα παιδιά είναι ορφανά και θα πρέπει ε, να στηρίζουμε τον ένα γονέα. Όταν όμως ε, έχουν και τους δύο γονείς τους τα παιδιά, το συμφέρον τους είναι να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε ας πούμε, την προσωπική βεντέτα και τις κόντρες που έχουν οι γονείς ε, και κρατάει χρόνια πολλές φορές. Και εγώ πολλές φορές πριν γίνω πολιτικός, πριν από πολλά χρόνια, έκανα τέτοια διαμεσολάβηση και ήμουν συζυγικός σύμβουλος και θα ήταν χρήσιμο αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει, δεν το ζητάω, δεν ζητάω να μου απαντήσετε, απλώ θα ήταν ενδιαφέρον για τους συναδέλφους να μάθουν αν δοκιμάσατε και αυτό. Yes, we was Ναι, δοκιμάσαμε. Το 2011 με διαμεσολαβητή του Κοινοβουλίου ε, για θέματα ε, παιδικής, απαγωγής παιδιών από γονέα αλλά υπήρχε μια κόκκινη γραμμή που ήταν η παρανομία. Η γυναίκα μου που ήταν αλλοδαπή ζήτησε να αναγνωριστεί το διαζύγιο και ε, de facto μια απόφαση ε, δικαστηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, απόφαση που πριν από τρεις μήνες είχε ακυρώσει το ελληνικό δικαστήριο λόγω παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οποιοδήποτε φιλικός διακανονισμός και επίλυση διαφοράς θα πρέπει να κινείται πάντα στα πλαίσια του νόμου. Δεύτερον, εγώ δεν ζητάω από το Κοινοβούλιο να δικάσει την υπόθεσή μου. Αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου. Να ζητήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά την ε, κείμενη νομοθεσία και το κράτο δικαίου και να εξηγήσω για την απόφαση αυτή για τα διαβατήρια. Όπω είπατε, να απόκειται στα κράτη-μέλη αυτό και στι αρμόδιε κρατικέ αρχέ να εκδίδουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Αλλά ο κανονισμό Βρυξέλλε 2 ισχύει από το 2005 και έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη, ε, με εξαίρεση τη Δανία. Δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν ε, για τον κανονισμό αυτό που λέει ξεκάθαρα ότι όταν έχεις γονική ευθύνη και μέρημνα παίρνεις και κρίσιμες αποφάσεις για το πού θα σπουδάσουν τα παιδιά σου, σε ποιο σχολείο θα πάνε, σε ποια χώρα θα ζουν κτλ. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των γονέων, τότε μπορεί το δικαστήριο να αποφασίσει του κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία. Αυτή είναι η απόφαση και αυτά ορίζει η απόφαση και συμφωνώ με την ε, κυρία Λεωνόρα Εύη αφού υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές με τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να γίνει μια σωστή ανάλυση του θέματος και της απόφασης αυτής για να καταλάβουμε πραγματικά τι ε, αποφαίνεται. Ευχαριστώ. Δεν είναι πολύ απλή αυτή η περίπτωση για να συνοψίσουμε. Μακάρι να ήταν, αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε, έχει και μια ανθρώπινη διάσταση. Σε κάποια στιγμή, χαίρομαι που το έθεσαν και κάποιοι συνάδελφοι. Εδώ γίνεται λόγος για παιδιά. 12 και 15, αν δεν απατώμε, έτσι. Α, 11 και 15 των. Είναι ακόμα παιδιά νεαρά παιδιά, ανήλικα. Είναι σε μια τρυφερή ηλικία, ευαίσθητη ηλικία που χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. Δηλαδή και πάλι θα σας παρακαλούσα, θα σας εκλυπαρούσα, κοιτάξτε το, προσπαθήστε να δείτε τι μπορεί να γίνει και θα ήθελα να επανέλθετε εσείς στη γραμματεία. Ξέρω ότι έχετε τώρα μια μακρά σχέση διαρκείας με τη γραμματεία για αυτό το θέμα ε, να εξηγήσετε αν προσπαθήσατε να κάνετε ένα διακανονισμό φιλικό προς το συμφέρον των παιδιών σας. Όχι για να συνεχιστεί αυτή η βεντέτα με την πρώην σύζυγό σας, να προσπαθήσετε να βρείτε μια λύση ε, για το συμφέρον των παιδιών, το καλό Δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι έχω δει πολλά, έχω ζήσει πολλά, έχω δει περιπτώσεις πολύ πιο ακραίες από αυτές που μας παρουσιάσετε και ακόμα εκεί δεν χρειάζεται δικαστήριο, δεν χρειάζεται να μιλήσετε. Απλώς σας λέω ότι χρησιμοποιώ το προνόμιο μου ως πρόεδρος αυτή τη στιγμή και επανέρχομαι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα εμείς, συνάδελφοι. Πρώτο, κάποιος, είπε, κάποιος συνάδελφος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και τίνω να συμφωνήσω. Παρ' όλα αυτά, είπαν οι συνάδελφοι ότι είναι πρόθυμοι να παρακολουθήσουν, να συνεχίσουν αυτή την υπόθεση, να το κοιτάξουν από άλλη σκοπιά και εγώ θα πρέπει να το λάβω σοβαρά υπόψη, αλλά θέλω να υπογραμμίσω και να το σημειώσετε όλοι παρακαλώ ότι Κύριε Γιαννόπουλε, δεν μπορούμε να σας δώσουμε φρούδες ελπίδες και προσδοκίες αυτό το θέμα από ε, σκοπιάς είναι μια υπόθεση όπου δεν μπορούμε να σας δώσουμε φρούδες, ελπίδες και ψευδεστήσεις. Βέβαια είναι στα χέρια σας να βρείτε τρόπο δικαστικό να το λύσετε και στα δικά μας να κάνουμε αυτό που ζήτησαν οι συνάδελφοι ως Επιτροπή. Δηλαδή, τα έξις. Να στείλουμε επιστολή στη Eurojust και να έχουμε ε, γραπτή ενημέρωση για το τι συμβαίνει, τι έχουν κάνει εκεί και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, γραπτή ανάλυση, ακόμα και αν πρέπει να σας πω ότι η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ καλή, μας εξήγησε με παραθέσεις και τα γεγονότα και τις αποφάσεις. Πάντως θα ήταν καλό να ε, έχουμε και γραπτό στην ανάλυση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να ανατρέξουμε και να επανέλθουμε και να την επικαλούμαστε. Στη συνέχεια θα στείλουμε επιστολή ε, στον Κύπριο Γενικό Εισαγγελέα και στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου και τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας. Και τελευταίο, χωρίς αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό βεβαίως, αφού έχουμε ομάδα εργασίας για θέματα ευημερία των παιδιών, η κυρία Πρόεδρος, κυρία Εύη. Κυρία Εύη, με χαρά θα το παραπέψω σε εσά και στην ομάδα εργασίας. So take, take it, the ball Παρακαλώ. Το μπαλάκι λοιπόν είναι στο γήπεδο της ομάδας εργασίας. Κάντε ό,τι μπορείτε, ό,τι περνάει από τα χέρια σας για να το εξετάσετε και από άλλη μια σκοπιά. Συμφωνούμε. Συνάδελφοι, συμφωνείτε με τα όσα πρότεινα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που σας έδωσα το λόγο προηγουμένως, δεν χρειάζεται να ξαναμιλήσετε, δεν πιστεύω. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που ήρθατε και εμείς έτσι θα προχωρήσουμε. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία και ίσως του χρόνου θα δούμε. Θα δούμε. Ελπίζομαι. Ευχαριστώ. Let's now move on to the next petition, which is item 12 on the agenda. Να περάσουμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, στην επόμενη αναφορά. ένας ε, πολίτης γερμανικής εισαγένειας ε, όσον αφορά την εφαρμογή δικαστικής απόφασης ώστε να του επιτρέπεται να ασκεί το δικαίωμά του να επισκέπτεται το παιδί του. Είναι εδώ ο αναφέρον. Θα ήθελα να του δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Γεια σας. Στα αγγλικά. Θα έρθω στο θέμα αυτό. Έχει απάγει το παιδί μου, η γυναίκα μου, η μητέρα του προς το Ηνωμένο Βασίλειο και έκτοτε δεν έχουμε επαφή καμία και καμία επικοινωνία. Βλέπετε ε, ε, στην οθόνη εδώ τι έχει γίνει από τη γέννηση του παιδιού. Πριν πω σε είναι τι που έχω να κάνω. Όταν έγινε συζήτηση για ένα παιδί που δεν θέλει να πάει στο σχολείο, αυτά τα θέματα δεν είναι κοινά, δεν είναι θέματα ε, που συζήτηση. είναι υποχρεωμένο το παιδί να πάει στο σχολείο. Δεν ρωτάς το παιδί και όταν αρχίσει και το ρωτάς αν θέλει όχι να δει ένα γονέα, ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Ιδιαίτερα ε, μπορεί να επηρεάζει ο ένας γονέας το παιδί ή κάποιος άλλος. επανέρχομαι λοιπόν στο παιδί μου. Την περασμένη φορά τα σταματήσαμε. Ε, υπήρξε απόφαση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει μια επιστολή μάλλον η Επιτροπή σας να στείλει επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό από ό,τι ξέρω. Το παιδί μου γεννήθηκε το 2004 και γύρω στο 2007 ήμασταν ήδη στα δικαστήρια, προσπαθήσαμε να το κάνουμε πολιτισμένα και ε, τα δικαστήρια της Μάλτας έβαλαν κοινωνικούς λειτουργούς και τα λοιπά. Ε, όχι, δεν ήταν ε, ο πατέρας επικίνδυνος. Ο πατέρας ερχόταν από τη Γερμανία, έβλεπε το παιδί του. το 2009 το έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα χρόνο το παιδί η μητέρα προσωρινά και αμέσως μετά την έλευση του παιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο χάθηκε η επαφή με... και τέσσερις μήνες έκανα για να βρω το παιδί μου. Και τότε υπήρξε ο κανονισμός ε, Βρυξέλλες 2α και ε, το 2010 με ενημέρωσαν γραπτός, αλλά και εγώ προσωπικά ενημέρωσα γραπτός και στη συνέχεια προσωπικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχω επαφή. Κοιτάξτε, εγώ δικηγόρος δεν είμαι και ιδιαίτερα τότε δεν τα ήξερα καθόλου αυτά τα νομικά ζητήματα. Και τελικά τι ανακάλυψα τότε. Βρέθηκε η μητέρα, πήρα ένα λογαριασμό μου, στείλαν 18.000 ε, λίρες Ε, για να βρω το παιδί μου. Σταμάτησα μετά από τρεις μήνες γιατί δεν μπορούσα να πληρώσω, γιατί αυτοί το έχουν κάνει μπίζνα εκεί πέρα. Ε, αργότερα, το 2010, α, εντωμεταξύ η μητέρα δεν μπορούσε να κρατήσει το παιδί πια στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είχε λήξει η δυνατότητα και το 2011 Ε, το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να το πάρω το παιδί μου και ε, να το βγάλω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν η τελευταία δυνατότητα να δω το παιδί μου και το παιδί φυσικά δεν θέλει να το παίρνει ο πατέρας του από το σχολείο και να το πηγαίνει σε άλλη χώρα. Το 2011 είχαμε δεύτερη απαγωγή, δηλαδή η μητέρα και πάλι πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν επέστρεψε και δεν ε, ε, εφαρμοζόταν σωστά ο νόμος, δηλαδή Βρυξέλλες 2 και ε, η, η Μαλτέζικη απόφαση ότι είχα τη δυνατότητα πέντε μέρες και μία νύχτα να βλέπω το παιδί μου. Το 2013 το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε μια απόφαση αλλά η Μάλτα διαφωνούσε, τελικά αποφάσισε δικαστήριο Βρετανικό και το 2015 και τώρα εκεί βρισκόμαστε ε, και τώρα έχω μάθει πώς έπρεπε να είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία, το Ηνωμένο Βασιλείο απέρριψε το αίτημά μου ε, για προδικαστικό ερώτημα στο Λουξεμβούργο, στο δικαστήριο, ε, που δεν είχε εκπνεύσει η προθεσμία, ήταν μια διετία. Το 2013 όταν πήρε απόφαση λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο, όρισαν ένα ψυχολόγο και επέστρεψε αυτή μια στιγμή γιατί τα έχω κάπως χάσει. Uh, λοιπόν, ορίστηκε ψυχολόγος, ειδικό για το παιδί και μετά από ένα χρόνο δεν υπήρξε πρόοδος, μετά ε, ξαναπήγα στα δικαστήρια και, και λέω «Παιδιά, δεν μπορώ να βλέπω το παιδί μου κάθε τρεις μήνες μία ώρα όταν έρχομαι στο Λονδίνο». Δεν έγινε τίποτα και το 2015 προσπάθησα να ξεφορτωθώ αυτό το δικαστή και ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, γιατί από το 2013 ήταν η ίδιος δικαστής δικαστήνα κιόλα που δεν ε, βοηθούσε να συναντάω το παιδί μου. Και μετά, όταν έμαθα τι γινόταν, ζήτησα να πάει στο Λουξεμβούργο, ακόμα και αν ήταν αργά, για προδικαστικό ερώτημα ως προς την ερμηνεία για το πώς επιβάλλεται ε, ο κανονισμός Βρυξέλλης 2α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι αυτό απαραίτητο κάθε φορά. Τι έκανε η Κομισιόν τώρα. Έχω σοβαρά ερωτηματικά ε, στην πολιτική αυτή για, για τη δικαιοσύνη. Η αστική δικαιοσύνη θα πρέπει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι θέμα πολιτικής αυτό, δεν είναι νομικά ζητήματα. Κάτι άλλο που ε, παρατήρησα πολύ προσεκτικά ήταν η υπόθεση του Μαξ Σερν στο δικαστήριο για το Safe Harbor. Είναι ήρωας πραγματικά, δικαιώθηκε. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνεί το ότι ήταν παραβίαση και κατάφερε να το φέρει στο δικαστήριο και να κερδίσει. Και ε, παρόλο που έχει το μονοπόλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κέρδισε, δικαιώθηκε στο δικαστήριο και το απάντησαν ότι όντω υπήρχε παραβίαση και είχε λάθος. Ε, Ήτανε, ε, είχε άδικο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Safe Harbor. Τώρα αυτό τι σημαίνει. Εγώ έχω ακόμα τη γονική μέρημνα και επιμέλεια και θέλω να έχω άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με το παιδί μου και θα πρότεινα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται ότι υπάρχει παραβίαση ε, Υπάρχει αυτό που λέγεται parental root cutting που κόβουν τους διάβλους επικοινωνίας. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα και χρειάζεται προδικαστικό ερώτημα και απόφαση για το, ε, από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου για την ερμηνεία πώς θα πρέπει να βλέπει ένας γονέας το παιδί του. Υπάρχει χάρτη σε θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπαίνει εδώ στην υπόθεση. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για διεθνές δίκαιο. Ίσως καλό θα ήταν να ε, βάλουμε και το χέρι στην τσέπη και να φέρουμε στο δικαστήριο αυτά τα θέματα. Είναι σχετική και η περίπτωσή μου και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, πηγαίνει στο δικαστήριο, πηγαίνει η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Currently και πρόκειται για αναθεώρηση τώρα του κανονισμού Βρυξέλλες 2α, αλλά δεν έχουμε καμιά ενημέρωση, δεν υπάρχει κανείς εξωτερικός εγώ ρώτησα, μπορώ να συμμετέχω εγώ ή κάποιος από το κοινοβούλιο σε αυτές τις συνεδριάσεις στις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Καμία ενημέρωση. Και τελικά έχουμε αυτή την υπόθεση, τη δική μου και την προηγούμενη του κυρίου Γιαννόπουλου. Δεν θα μπορούσαμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, Βρυξέλλες 2, να τις αφήσουμε ανοιχτές μέχρι να έρθει νέα πρόταση και να κοιτάξουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα και αν εφαρμόζεται σωστά ο, δρόμ, ο νόμος. Συγγνώμη. Sorry που μακρηγόρησα. Thank you very much. And yes, we are running short. Ναι, πράγματι, έχει περάσει ο χρόνος, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γκρούμπισιτς και πάλι, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον αναφέροντα. Θα μπορούσα να είμαι σύντομο νομίζω, γιατί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αποστείλει περίπου 20 επιστολές ε, στον αναφέροντα, όπω επίση έχει απαντήσει και σε 30 αιτήματα πρόσβαση σε έγγραφα και η αναφορά αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζει τίποτε το καινούριο που να μην έχει εξετάσει από κοινού με την νομική υπηρεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νόημα όλης αυτής της καταγγελίας αφορά τον κανονισμό ε, Βρυξέλλες 2 ειδικότερα όσον αφορά την επιβολή της ε, μαλτέζικης απόφασης ε, των δικαιωμάτων επίσκεψης του αναφέροντος στο παιδί του Δυστυχώς ε, έχουμε πολλές φορές πει στον αναφέροντα, πολλές φορές ότι οι Βρυξέλλες 2α ορίζουν ε, πώς μία απόφαση σαν αυτήν της Μάλτας σε σχέση με τα δικαιώματα επίσκεψης ε, αναφέρει μόνο πώς μπορεί να αναγνωριστεί και πώς μπορεί να επιβληθεί σε κάποιο κράτος μέλος. Όταν όμως πρόκειται για την επιβολή στο κράτος μέλος, ε, ο κανονισμός λέει κατακάθαρα ότι η πραγματική εφαρμογή, ε, πώς ακριβώς πρέπει να γίνει λοιπόν η διαδικασία της εφαρμογής, επαφίεται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους. Η Βρυξέλλες 2α είναι ένα... Ε, ε, μέσω ιδιωτικού διεθνούς δικαίου γνωρίζουμε ότι ήρθαν σε επαφή τα Βρετανικά δικαστήρια με τον αναφέροντα και του εξήγησαν ποιο είναι το πρόβλημα στη διαδικασία της ε, επιβολής ε, της εφαρμογής απόφασης αυτής και η... επειδή ο ίδιος ο αναφέρον έχει όπως ε, έχουμε πει πολλές φορές τον αναφέροντα, ε, επειδή έχει, περάσει πολύ καιρό ήδη που έχει πάει η ε, γυναίκα του με το παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει του άρθρου 10 τα Βρετανικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μόνο αυτά τα στοιχεία μπορεί να λάβει υπόψη γιατί όπως σας είπα ο κανονισμός είναι ένα μέσο ιδιωτικού διεθνούς δικαίου δεν έχουμε δυστυχώς καμία άλλη δικαιοδοσία ως ως προς το να επιβάλλουμε την εφαρμογή της απόφασης και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει έρθει σε επαφή ακόμη με το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δεν μπορούμε να δούμε, ε, δεν μπορούμε να ε, διαπιστώσουμε παραβίωση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και μόνο σε περίπτωση παραβίασης ε, μπορεί ε, να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επαφή με το κράτος μέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, για τις επεξηγήσεις σας. Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Θα δώσω και πάλι το λόγο στον αναφέροντα για ένα λεπτό γιατί προηγουμένως μιλήσατε ε, πολύ περισσότερο. Καλώς. Θα επανέλθω στο πρώτο σημείο, διότι αποφαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βαρεθεί τα διαγράμματά μου. Ε, ζητώ ενημέρωση. Ζητώ από τον Ευρωπαίο ε, Διαμεσολαβητή ήδη από το 2013 να επιληφθεί. Ζητώ και οδηγίες πώς να προχωρήσω και τίποτα δεν έγινε. Τι να κάνω στο Ενωμένο Βασίλειο όταν ε, ήξερα ότι αυτοί θα το πηγαίνουν στα δικαστήρια. Τώρα Ξέρω τώρα όμως το γνωρίζω αυτό ότι έπρεπε να είχαμε ρωτήσει το Λουξεμβούργο για προδικαστικό ερώτημα και αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση δικαιοσύνη, δεν είναι δική τη δουλειά. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή πρέπει να το κοιτάξει. Νομίζω ότι είναι λάθο η απάντηση. Δεύτερον, ζήτησα ε, επίσημα επίση. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, να ληφθεί υπόψη αυτό στα Βρετανικά δικαστήρια. Αυτοί το απέρριψαν ω αβάσιμο. Είπα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται και μου λένε ότι όχι. Ε, ο Μαξ Ρέμ όμως λέει στο βίντεο του ότι είναι πάγια τακτική αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Εκλαμβάνω ότι ζητήσατε το λόγο. Θέλατε το λόγο και αποσυρθήκατε ή θέλετε το λόγο τελικά. Θέλετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Ήθελα να πω ότι θα ήθελα να παραμείνει η αναφορά αυτή ανοιχτή, ούτω ώστε να γίνει μια περαιτέρω εις βάθος ανάλυση στην ομάδα εργασίας του χρόνου. Για να διευκρινίσουμε όλα τα ζητήματα που έθεσε ο αναφέρον, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, είναι συγκεκριμένη η κατάσταση. Χρειάζομαι περισσότερη ανάλυση των θεμάτων. Και κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια υπόθεση όπου οι Βρυξέλλες 2 δεν έχουν εφαρμοστεί από το κράτος ε, μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε να υπάρχει λαθασμένη εφαρμογή του Βρυξέλλες 2. Διότι κάθε φορά με τον κανονισμό αυτό Βρυξέλλες 2 βλέπουμε είτε εφαρμόζεται είτε με κάποιο, εφαρμόζεται με κάποιο τρόπο ανεπαρκή. Φαύλος κύκλος γίνεται. Αυτό αισθάνομαι. Ας κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Για να μπούμε εις βάθος τους επόμενους. Να σας πω την αλήθεια, λέει ο Πρόεδρος, το να παραμείνει ανοιχτή αναφορά όταν είναι εδώ, έχει έρθει ο αναφέρον τρεις φορές και 20 φορές έχει λάβει γραπτές απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να διατηρούμε ένα φαύλο κύκλο κατά την άποψή μου και να δημιουργούμε ψεύτικες προσδοκίες. Αν αισθάνεστε, αν ότι κινείστε σε φαύλο κύκλο, σπάστε τον κύκλο. Ε, κυρία Πιτέλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πράγματι. Κινούμαστε σε ένα φαυλοκύκλο και δεν βρίσκουν τη διέξοδο οι ε, διάφοροι αρμόδιοι. Οι υιοθεσίε και συναφή θέματα είναι δυσχερέστατα νομικά προβλήματα. Στην περίπτωση διαφοράς μεταξύ των γονέων δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο κάποιος αξιωματούχος μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Τι να κάνουν, να πάρουν το παιδί από τους γονείς, ένας γονέας δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του άλλου γονιού. Το να επιτευχθεί συνένεση μεταξύ δύο ανθρώπων ενός διαζευμένου ζευγαριού δεν είναι κάτι που το αναλαμβάνουν οι διάφοροι αξιωματούχοι. Είναι κάτι για τους, που αφορά τους ψυχολόγους, τους μεσολαβητές και καμιά φορά και αυτοί δεν καταφέρουν να βρουν λύση. Διερωτώ λοιπόν, πώς να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Μπορούν οι γονείς να υποχρεωθούν να συμφωνήσουν από κάποιον αξιωματούχο που θα κινηθεί με κάποιον αυταρχικό τρόπο. Μπορεί να το πετύχει αυτό κάποιο δικαστήριο. Δεν νομίζω. Υποκρινόμαστε. Κάνουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Θα παραμείνει άλλη μία ακόμα αναφορά ανοιχτή μέχρι ότου ενηλικιωθεί το παιδί και ίσως όταν είναι ενήλικες τα παιδιά θα αποκτήσουν καλές σχέσεις με τον ένα γονιό και με τους δύο γονείς ή θα μισούν και τους δύο γονείς. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η εμπειρία μας μας δίνει τη δυνατότητα, μας δείχνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πιτέλα, λέει πρόεδρος. Τώρα πώς να συνοψίσω το όλο θέμα. Θα ήθελα να πω έτσι πραγματικά ότι να κρατήσουμε αυτή την αφορά ανοιχτή δεν είναι προς όφελος, προς συμφέρον της Επιτροπής μας. Ήρθατε εδώ, κύριε μου, τρεις φορές ήδη. Οι ανταλλαγές και συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίστηκαν επανειλημμένα. 20 επιστολές ανταλλάχθησαν. Πιθανότατα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα εμείς σαν Επιτροπή. Και ξανά, Θέλω να πω ότι δεν θέλω να δημιουργώ ψευδείς προσδοκίες. Έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημά σας. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή. Η κυρία Εύη, από ό,τι άκουσα, θα επιθυμούσε να κινηθεί. Αλλά δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες ε, ε, πληροφορίες να εξεταστούν. Αλλά θα μπορούσαμε να κλείσουμε την αναφορά και να το παραπέμψουμε το θέμα στην ομάδα εργασίας, αν θέλετε να ασχοληθείτε με το θέμα. Αυτή είναι μια πρόταση. Και κλείνουμε την αναφορά. Την κλείνουμε και σαν ενημερωτικό, σαν ενημερωτική υπόθεση μπορεί να συζητηθεί το θέμα στα πλαίσια που άπτονται των παιδικών θεμάτων, σαν κάτι πρόσθετο. Όχι ε, να ξανανοίξει η αναφορά, αλλά να το έχετε σαν σημείο αναφορά, σαν υπόθεση αναφοράς. Είναι μια δυνατότητα. Κυρία μου, σα έδωσα ήδη το λόγο. Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι, στρέφομαι προς τους συναδέλφους. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ναι, από ό,τι βλέπω, γνέφουν. Η κυρία Σντανόκα. Κοιτάξτε Πρόεδρε, κατανοώ, κατανοώ, το καταλαβαίνω, ότι το συζητήσαμε. Σήμερα είπαμε ότι χρειάζεται καλύτερος ορισμός του συνήθους τόπου διαμονής, habitual residence, συγγνώμη. Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τις Βρυξέλλες 2, τι να πω, θα ήταν καλύτερο να μην δίνουμε ψευδείς υποσχέσεις, αλλά θα ήθελα να παραμείνει αναφορά. Μπορούμε να αποδείξουμε ως επιχείρημα ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα. Ξέρουμε αρκετές υποθέσεις που αφορούν τη Βρετανία και το πρόβλημα έγκυται στο ότι δεν μπορεί να οριστεί ο συνήθις τόπος διαμονής χωρίς ψευδείς υποσχέσεις να αφήσουμε το θέμα συζητηθεί στα πλαίσια της συζητήσεως της Ολομελίας για, το, τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 να παραμείνει ανοιχτή υπόθεση. Είμαι και εγώ μέλος της ομάδας εργασίας και θα ήθελα να το εξετάσουμε. να, όταν γίνουν οι συζητήσεις στην ομάδα εργασίας ήταν καλύτερο να εκκρεμεί ακόμα, να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η υπόθεση. Η λύση σας ενδεχομένως είναι η καλύτερη. Βάσει των όσων ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εσά τον αναφέροντα και γνωρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση, θα ήταν δίκιο και καλό. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Πετήρα να μην δημιουργούμε ψευδείς προσδοκίες και ελπίδες. Όλες οι αναφορές που έχουν υποβληθεί όλα αυτά τα χρόνια που αφορούσαν το πώς αντιμετωπίζονται οι υποθέσεις της Ασίας των παιδιών στην Ηνωμένο Βασίλειο θα, είναι, θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της Επιτροπής θα δούμε τι θα γίνει με επίσκεψη στο Λονδίνο και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε μία ανάδραση του τρόπο. Στο να παραμείνει ανοιχτή αναφορά όμως θεωρώ ότι δημιουργεί ψευδείς ελπίδες και ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να βρει λύση. Πέρα το ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε μια διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής που θα έπρεπε να είναι και ο στόχος μας. Ευχαριστώ πολύ. Μπεατρίς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω μόνο ότι συμφωνώ με την πρότασή σας Πιστεύω ότι η ειλικρίνεια και η τιμιότητα της Επιτροπής μας εκεί ε, δράζεται. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι. Από την αρχή δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, ε, με τους ανηλίκους, όπως είπε η συνάδελφος. Ε, τώρα συζητάμε την επίσκεψη στο Λονδίνο και τα συμπεράσματα και σε κάθε πολιτική ομάδα τα παιδιά και ό,τι έχουν να κάνουν με παιδιά και διαδικασίες που δεν έχουν να κάνουν με την ε, πρόνοια και την ευημερία των παιδιών. Τώρα να αφήσουμε ανοιχτή ή όχι την ε, αναφορά αυτή. Να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε Βέβαια δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν θα συνεχίσει να δουλεύει για την πρόθεση της νομοθεσίας. Αλλά αυτή η αναφορά έχει κάνει το κύκλο της, έχει κλείσει και τώρα πραγματικά κυνηγάει την ουρά της ένα φαύλο κύκλο. Ε, είναι πολύ ε, έντιμο και πολύ σωστό και πολύ μεγάλη κατανόηση δείχνει πρόεδρος αυτό που προτείνει. Ευχαριστώ. Η κυρία Πιτέρα. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Τα παιδιά είναι δυστυχισμένα γιατί δεν γνωρίζουμε εάν τα παιδιά που διαμένουν με τη μητέρα τους είναι ευτυχισμένα ή δυστυχισμένα. Δεν ξέρουμε τη δική τους ε, άποψη. Εμένα θα με ενδιέφερε κατά πόσο ε, βρίσκονται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να ε, μεγαλώσουν φυσιολογικά, είναι υγιεί, έχουν τρόφιμα, εκπαίδευση ε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να χρήζει επιστημονικής καθοδήγησης. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν ε, διαφωνίες. Ε, θέλουμε λοιπόν να... Θα ήθελα να ξέρω πώς νιώθουν τα παιδιά γι' αυτό. Να κάνουμε λοιπόν την εξή ερώτηση. Οι κοινωνικές υπηρεσίε γνωρίζουν κατά πόσο τα παιδιά λαμβάνουν σωστή φροντίδα. Γιατί εγώ δεν θα ήθελα να μπαίνω στη μέση μίας διαφωνίας μεταξύ δύο ενηλίκων. Με ενδιαφέρουν ε, τα παιδιά πώς νιώθουν, γιατί έχουν ε, πολύ σημαντικά ε, δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό που είπατε είναι ακριβώς το βασικό πράγμα. Η ευημερία των παιδιών. Άκουσα όλους τους συναδέλφους και νομίζω ότι μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Αρχικά είχα την προώθηση να κλείσω την αναφορά αυτή. Άλλωστε έχει έρθει τρεις φορές εδώ αναφέρον και όπως είπα ήμασταν διεξοδικότατοι. Δεν υπάρχει κανένα άλλη μαγική λύση που να μπορούμε να βρούμε. Έχοντας όμως ακούσει τους συναδέλφους νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να την κλείσουμε την αναφορά αλλά αφού την κλείσουμε να την στείλουμε στην ομάδα εργασίας ε, για τα θέματα των παιδιών για περισσότερη συζήτηση και εξέταση όταν, ε, να, ληφθεί υπόψη δηλαδή όταν ε, θα υπάρξει έκθεση από την ομάδα εργασίας, η Λεωνόρα. Να προσθέσω απλώς ότι δεν συμφωνώ με αυτό που είπε η συνάδελφος Πιτέρα για τον απλούστατο λόγο που είναι εξή. Δεν μπορούμε εμείς να διερευνήσουμε το όλο θέμα, να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι ανήλικοι. Μπαίνουμε σε μια σφαίρα που δεν είναι στην αρμοδιότητά μας και εμείς είμαστε εδώ για να φροντίσουμε τόσο τα δικαιώματα και των δύο γονέων να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους γίνονται σεβαστά. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι προφανές ότι πρέπει να είναι σαφές ότι εδώ μιλάμε βέβαια για το καλό εκεί και το όφελος των παιδιών. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το πεδίο γιατί δεν εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα. Εγώ το ερμήνευσα εγώ την ε, παρέμβαση της κυρίας Πιτέρα. Θεώρησα ότι έδειξε ανθρώπινο ενδιαφέρον για το θέμα και θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό που βλέπουμε είναι μία πλευρά, μία όψη του νομίσματος. Έχουμε δύο γονείς σε αυτή την υπόθεση, είδαμε τη μία όψη του νομίσματος. Επανειλημμένα, δεν γνωρίζουμε τίποτα για τα παιδιά ούτε για τη μητέρα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη από όλους τους παρισταμένους. Λοιπόν, συνάδελφοι, να το κάνουμε αυτό. Να κλείσουμε την αναφορά τελικά. Και σαν σημείο αναφορά στο θέμα αναφορά θα προωθηθεί προ ενημέρωση και περαιτέρω συζητήσει στην ομάδα εργασία για την ευημερία των παιδιών. Ναι, ωραία. Καλώ αυτό θα κάνουμε. Σα ευχαριστώ πολύ και προ τον αναφέροντα πρέπει να σα πω ότι σα έχω δώσει ήδη το λόγο, λυπάμαι και έχουμε καθυστερήσει, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το θέμα. Ευχαριστώ του αναφέροντε που ήρθαν εδώ και τώρα είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε διότι προχωρούμε στο επόμενο σημείο της σα διάταξης που αφορά εντελώς διαφορετικό θέμα, αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, η 723 αναφορά του 2014 αυτή που συζητάμε. Αναφέρον εδώ η Ιωάννα Σβάμπε, είναι εδώ η αναφέρουσα, που έχει το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Thank you. As the... Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, επειδή το σκάνδαλο με το ελογίσιο κρέα σιγά σιγά φεύγει από τη μνήμη των Ευρωπαίων πολιτών και των πολιτικών, υπάρχει ένα ακόμη τέτοιο σκάνδαλο, το οποίο η Humane Society International θα ήθελε να αναφέρει σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο που συμπεριλαμβάνει ε, ενδεχόμενου κινδύνου για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και ένα σκάνδαλο για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε μπορεί να λύσει ταχύτατα. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα γιατί μου δίνει την ευκαιρία να συζητήσω ε, το θέμα αυτό που αντιμετωπίζει την ασφάλεια του κρέατος αλόγων που εισάγεται από, ε, ε, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο χιλιάδες τόνων κρέας, κρέατος αλόγων εισάγονται στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στις κάτω χώρες ή στην Ιταλία από τρίτες χώρες ε, το περισσότερο, το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του κρέατος προέρχεται από τη Βόρεια ή Νότια Αμερική, όπου οι, τα άλογα δεν θεωρούνται ότι μπορούν να παράγουν τρόφιμα ε, από το κρέα τους ε, ή το, ιστορικό τους, το ιστορικό των αλόγων αυτών δεν, δεν, δεν τα καθιστά κατάλληλα. Από τον Ιούλιο του 2010 το ιστορικό, το ιατρικό δείχνουν, δείχνει ότι ε, δεν έχουν γίνει σεβαστές οι περίοδοι ε, που θα έπρεπε να υπάρξουν πριν το σφαγιασμό των ζώων. Κάθε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να συμφωνεί με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαμονή των αλόγων και το σχέδιο επιτήρησης καταλήπων πριν από το σφαγιασμό. Στην αναφορά μας αναφέρουμε ακριβώς αυτό το γεγονός ε, έχουμε πάρα πολλές φορές ε, ακούσει ελέγχους ε, από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Από την υποβολή της αναφοράς μας τον Απρίλιο του 2014 και μετά από μακροχρόνια εκστρατεία και πίεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους απαγόρευσε την εισαγωγή του κρέατος αλόγων από το Μεξικό επειδή υπήρχαν σοβαρές ε, ε, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τη διεξαγωγή ελέγχων και τη χρήση των απαγορευμένων ουσιών, ε, κάτι που είχε φανεί σε ελέγχους από το Γραφείο Τροφίμων και Εκτινιατρικών Θεμάτων. Τέτοιου είδους προβλήματα ειχνημότητας υπάρχουν και με άλλες χώρες που εξάγουν όπως ο Καναδάς και η Αργεντινή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κατά τη γνώμη μας λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με, τον, με το Καναδά ε, δεκάδες χιλιάδες ε, ε, αμερικανικά άλογα μεταφέρονται στον Καναδά κάθε χρόνο για να σφαγιαστούν για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αμερικανικά άλογα είναι 70% όλων των αλόγων που σφαγιάζονται στον Καναδά για παραγωγή κρέατος. Τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον τελευταίο της ε, έλεγχο σε σχέση με τον ε, Καναδά. Πολύ μεγάλες ανησυχίες υπήρχαν σε σχέση με την αξιοπιστία των αλόγων ε, και για τα καναδικά και για τα αμερικανικά άλογα που προορίζονταν για εξαγωγές κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως ο οργανισμός μας έχει πολλές φορές διαπιστώσει, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι δεν έχει χορηγηθεί απαγορευμένη ουσία στα ζώα αυτά ανταποκρινόμενη σε μία πρόσφατη διακομματική κοινοβουλευτική ερώτηση, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στο πρόγραμμά της για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Τα μέτρα που προτάθηκαν ε, συμπεριλαμβάνουν την τροποποίηση του πιστοποιητικού εισαγωγής, την ύπαρξη ισοδυναμίας απαιτήσεων σε σχέση με τις ε, εκτινιατρικές θεραπείες στον Καναδά και επίσης υποχρεωτική διαμονή έξι μηνών για τα άλογα η χώρα σφαγιασμού. Όμως ε, το να υπάρξει κάτι τέτοιο ε, δεν θα παρεμποδίσει το γεγονός ότι κάποια άλογα στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευμένες ουσίες ε, να, από το, να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως να κινδυνεύσουν Ευρωπαίοι πολίτες, η υγεία Ευρωπαίων πολιτών οι ε, ουσίες αυτές αν αν, που, που αν χρησιμοποιηθούν σε ε, άλογα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται απαγορευμένες, ε, δεν είναι απαγορευμένο να χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένε Πολιτείες. Εμεί πιστεύουμε ότι τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα λύσουν το πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα τη ασφάλεια τροφίμων, ούτε τη συχνηλασιμότητα. Και βεβαίω θα δημιουργήσει προβλήματα υγεία και ευημερία. Σε σχέση με την Αργεντινή, παρά το γεγονό ότι ο έλεγχο του FVO ανέφερε ότι η κατάσταση είναι γενικά ικανοποιητική. Μια καθυστερημένη εισαγωγή η υποχρεωτική θεραπείας του ιστορικού των υποειδών και ε, αποδεκτικών στοιχείων ότι δεν έχουν χειρουργηθεί απαγορευμένες ε, ε ουσίες υπονομεύει την αξιοπιστία ε, των εξαγωγών σε σχέση με το κρέας των ζώων αυτών. Στην Αργεντινή ε, κυρίως οι φενιλβουταζόνη και τα αντιπαρασιτικά μπορούν να αγοραστούν χωρίς συνταγή Όμω, οι ελεγκτές του FVO ε, αναγνώρισαν ότι τέτοιου είδου ουσίε χρησιμοποιούνται σε αγροτικέ εκμεταλλεύσεις ε, που ε, έχουν παράσχει άλογα σε κέντρα συλλογή για σφαγιασμό. Όσον αφορά τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε η επόμενη έκθεση του Γραφείου Τροφίμων και Εκτινιατρικών που αναμενόταν για αυτή τη χρονιά θα δημοσιευθεί. Και ολοκληρώνοντας, επειδή δεν έχω χρόνο, είναι σαφές ε, για μας ε, ότι η ασφάλεια του κρέατος αυτού που εισάγεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι πολύ ε, αμφισβητήσιμη και ζητούμε από την Επιτροπή Αναφορών να αναλυφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εισαγωγές αλογίσιου κρέατος από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανασταλούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And since... Ευχαριστώ πολύ. Ο αναφέρω να απουσιάζει η πορτογαλική ε, οργάνωση, αλλά η απάντηση είναι η ίδια και για τους δύο, γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή <laughs> Επιτροπή, ε, ιδιαίτερα ε, στον κύριο Μπλούμενταλ. Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε. <coughs> Ευχαριστώ τη δόκτωρα Σφάπ για την παρουσίαση της αναφοράς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, ε, εξονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οργάνωσή της για όλα όσα κάνει για την ευημερία των υποειδών. Το θέμα είναι πάρα πολύ τεχνικό. Να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή στους ε, τρέχοντες κανόνες και διαδικασίες εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις εισαγωγές κρέατος. Όπως γνωρίζετε όλοι, έχουμε εναρμονισμένους κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και την ευημερία των ζώων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή μπορούν να κυκλοφορούν τα αγαθά ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή συσταχθούν, έχουν πρόσβαση και στα 28 κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους κανόνες γενικά. Γενικά τα εισαγόμενα προϊόντα και το κρέας θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στα πρότυπά τους. Οι αρμόδιες αρχές των εξαγωγικών ε, κρατών που εξάγουν τρόφιμα δηλαδή θα πρέπει να πιστοποιούν και να εγγυούνται την τήρηση των κανόνων με ε, επίσημα πιστοποιητικά. Επιπλέον, όταν εισάγεται ποσότητα κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κρεοσκοπικοί έλεγχοι στα σύνορα με επίσημους ε, επιθεωρητές που ελέγχουν εάν και κατά πόσο τηρούνται όλα τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προδιαγραφές τα κατάλοιπα από φάρμακα, η ύπαρξή τους ή η αποσια τους, είναι κάτι που θα πρέπει να ελέγχουν οι τρίτες χώρες πριν την εξαγωγή ε, από ένα σύστημα το οποίο ελέγχει και εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, ε, οι ε, επιθεωρήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Γραφείου του Κτηνιατρικού που εδρεύει στο Grange ε, της Ιρλανδίας ε, ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν και τους κανόνες και την εφαρμογή τους. Το γραφείο για τα κτηνιατρικά και τα τρόφιμα ξέρετε ότι κάνει του ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να δώσει τα απαραίτητα χένια η τρίτη χώρα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσωπικά, ε, προσωρινά συγγνώμη, να απαγορεύσει το εμπόριο. Μέχρι να δείξει το κράτος ότι έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις και μπορεί και πάλι να φέρει τις εγγύσεις αυτές. Άλλη δυνατότητα είναι να ε, προτείνει συστάσεις στις τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να παρακολουθούν οι τρίτες χώρες και πάλι ελέγχει το Γραφείο Κτηνιατρικών και Τροφίμων. Για τον Καναδά ισχύει αυτό μέχρι τώρα. Έχουν γίνει έλεγχοι τα τελευταία χρόνια στον Καναδά από την υπηρεσία κτηνιατρικών και τροφίμων. Δεν έχει αποδειχθεί σοβαρός ε, υπαρκτός κίνδυνος για τις εξαγωγές υπείου κρέατος. Δηλαδή κρέας αλόγου αυτό. Ε, και δεν ε, έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε κτηνιατρική συμφωνία με τις καναδικές αρχές και υπό τις όρους συμφωνίας αυτής κάνουμε πολύ τακτικούς ε, ελέγχους, συνεδριάσεις, επικοινωνία. Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία για όλα τα θέματα και για την εξαγωγή κρέατος αλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το ίδιο το κρέας αυτό τώρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση και το σύστημα τα τελευταία χρόνια. Παρ' αυτά, όπως είπε και η δόκτωρ ΠΑΠ, η αρμόδια υπηρεσία τροφίμων και εκτινιατρικών, έκανε κάποιους ελέγχους που απέδειξαν ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιητική η κατάσταση στον Καναδά ακόμα. Άρα χρειάζεται ε, περαιτέρω σύστημα βελτίωση των εγγύσεων. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τροπολογίες ε, στα πιστοποιητικά εισαγωγής για το ε, ε, ήπιο κρέας και ε, όταν θα έχουμε αυτό το νέο πιστοποιητικό θα είμαστε βέβαιοι ότι θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και στις τρίτες χώρες με εκείνους που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να διαμένουν τα ζώα ζωντανά στη χώρα σφαγής τους για πάνω από έξι μήνες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που ε, επανειλημμένα λέγουν οι αναφέροντα ότι ε, πηγαίνουν στον Καναδά, τα σφάζουν σε 48 ώρες και εξάγουν το κρέα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μένουν 6 μήνες στον Καναδά <coughs> όπως ισχύει. Αυτές οι αλλαγέ λοιπόν στα πιστοποιητικά εισαγωγή ε, που ε, θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικές αλλαγέ. έχουν συζητηθεί με τα κράτη-μέλη και τώρα και σύμφωνα με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις τα αποστέλουμε στις εν λόγω τρίτες χώρες για να τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν τα σχόλιά τους uh, και περιμένουμε να εγκριθεί αυτό το νέο πιστοποιητικό στα αρχές του επομένου έτους και να αλλάξει ο τύπος ε, του πιστοποιητικού εισαγωγής και αυτό είναι πραγματική βελτίωση. Για την Αργεντινή τώρα, Έγινε και εκεί έλεγχος πέρσι από το γραφείο των ε, τροφίμων και κτηνιατρικών και τι βρήκανε, ότι παρά τις κάποιες αδυναμίες, το σύστημα ελέγχου της Αργεντινής δίνει τα χέγγια για την πιστοποίηση για τον οπό η ποιο κρέας που εξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη δεν είναι ακόμα έτοιμα τα απορίσματα και όταν ολοκληρωθούν και ε, τα σχολιάσουν οι τρίτες χώρες θα δημοσιευθούν. Thank you very much, Thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε συναδέλφους. Mrs. Hazekamp. κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους αναφέροντες που έθεσαν το ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια είχαν πολλά σκάνδαλα στον αφορά το λογίσιο κρέας. Δεν απειλήσαν μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά είναι καταστροφικά και για τα ζώα. Το κρέας αλόγων που έρχονται απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πωλείται το κρέας αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ συχνά βγαίνει από κατοικίδια άλογα και άλογα αγώνων. και έχουν υποστεί θεραπεία με φάρμακα τα οποία δεν επιτρέπονται στην ε, τροφική αλυσίδα. Μεταφέρθηκαν τα ζώα ζωντανά για αρκετές μέρες πριν φτάσουν στα σφαγεία και πολλά από αυτά ασθενούν ή πληγώνονται ή πολλά έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια των μεταφορών. Πάνω απ' όλα οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές αγνοούνται πολύ συχνά στα σφαγεία. Η κατανάλωση κρέατος ζώων είναι ένας κίνδυνος όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Κυρίως η πολλα εχουν πεθανει κατα διαρκεια των μεταφορων αλόγων είναι ένας κίνδυνος. Όπως είπα, πολύ συχνά δεν γνωρίζουμε την προέλευση των αλόγων αυτών. Και ο κίνδυνος είναι μεγάλος ότι έχουν πάρει φάρμακα που δεν θέλουμε να τα τρώμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά με τα αμερικανικά άλογα που μεταφέρονται στον Καναδά, μπορείτε να μας πείτε πότε η υποχρεωτική διαμονή ή εξάμεινος θα εφαρμοστεί. Δεν θα ήταν καλύτερο να αυτό ισχύσει όχι μόνο για τον Καναδά αλλά και για άλλες χώρες. Όλες τις χώρες στις οποίες σφαγιάζονται τα άλογα. Πώς θα λύσετε το πρόβλημα με το καναδέζικο κρέας το οποίο υπόκειται σε κατεργασία στη ΣΥΠΑ με ουσίες που δεν επιτρέπονται στην τροφική αλυσίδα και δεν μπορούμε να βρούμε ακριβώς εάν τηρούνται τα ε, ανώτατα όρια των καταλήπων. Τέλος, αντιμετωπίσαμε με πολλά σκάνδαλα όσον αφορά το αλογίσιο κρέα. Αλογίσιο κρέα που προερχόταν όχι μόνο απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων, αλλά κυρίω η υγεία και η ευημερία των αλόγων θα ωφεληθούν καλύτερα αν δεν εισάγουμε καθόλου αλογίσιο ε, κρέα και απαγορεύσουμε την πώληση στην Ευρώπη αλογίσιου κρέατος ανεξάρτητα από την προέλευση αυτού. Ευχαριστώ. Τζουντ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Οπότε από αυτά που μόλις ακούσαμε θα συνεχίσω κι εγώ. Τα τελευταία χρόνια η εμπιστοσύνη στην τροφική αλυσίδα και στον εφοδιασμό μας σε τρόφιμα έχει πληγεί τα μάλα από τα σκάνδαλα με το λογίσιο κρέας. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα που δεν νόμιζα ότι τρώμε πολύ αλογίσιο κρέα, Ανακαλύψαμε ότι το τρώγαμε, αλλά δεν το ξέραμε. Άρα υπάρχουν ε, σοβαρές ανησυχίες. Εγώ τα βλέπω κάπως διαφορετικά. Κοιτάζω περισσότερο τη δεύτερη αναφορά, όπου το θέμα συνδέεται περισσότερο με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και σε σχέση με τον Καναδά με την ε, γενική αυτή εμπορική συμφωνία που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο πιθανότατα του χρόνου προς ε, λήψη αποφάσεως. Αξίζει λοιπόν να το εξετάσουμε το θέμα. Να δούμε δηλαδή πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά αυτή την αναφορά. Λοιπόν, πάνω σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω κάτι. Ξεκινήσαμε ακούγοντα ότι ποτέ δεν υπήρχαν συστηματικά στοιχεία για προβλήματα στον Καναδά, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επέφεραν βελτιώσει οι Καναδοί, αλλά δεν είναι ακόμα ικανοποιητική κατάσταση. Διάβασα την έκθεση του, της υπηρεσίας, του ελέγχου που έγινε για θέματα κτηνιατρικά και για τρόφιμα του περασμένου Μαΐου. Η υπηρεσία, η αρμόδια, βρήκε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το λογίσιο κρέας. Άρα με προβληματίζει όλη η παρουσίαση του ζητήματος. Είναι καλό ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Είναι καλό ότι το πιστοποιητικό εισαγωγής έχει κάπως επικαιροποιηθεί. Αλλά έχουμε επαφές με τους Καναδούς και με τους Αμερικανούς και είναι σημαντικό να συζητούμε μαζί τους σύγκληση όσον αφορά τα αριθμιστικά θέματα, όσον αφορά τα θέματα φυτογενομικής προστασίας κλπ. Και, και πώς αυτά επηρεάζουν ε, τις εμπορικές μας σχέσεις. Όλα αυτά θα λάβουμε υπόψη και θα έλεγα να, τα, να παραπέψουμε αυτές τις αναφορές στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή Εμπορίου, Εξωτερικού Εμπορίου, διότι αυτά που συζητούμε εδώ επηρεάζουν αυτά που συζητούν οι άλλες επιτροπές και κυρίως την Επιτροπή Περιβάλλοντος μετά από το σκάνδαλο με το το θέμα της ανιχνευσιμότητας και στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου επίσης υπάρχει σχέση με τις συζητήσεις που διεξάγονται όσον αφορά τα πρότυπά μας για τις εμπορικές συμφωνίες και τα θέματα υγείας. Θα θέλαμε λεπτομερέστερες συζητήσεις. Έχουμε ομάδα εποπτείας στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου που εστιάζεται επί του Καναδά. Θα έπρεπε να ζητήσουμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής να τεθεί το συγκεκριμένο θέμα στην ε, ομάδα να δούμε τι διασυνδέσεις υπάρχουν μεταξύ αυτών που συζητάμε και του τρόπου με τον οποίο εκφράζονται οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΦΑΟ όταν διαπραγματευόμαστε τη συμφωνία και τι θα ακολουθήσει μετά τη σύναψη συμφωνίας. Αυτά έχω να πω λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καμιά φορά είναι καλό κανείς να προεδρεύει της Επιτροπής, γιατί βλέπει κανείς ότι έχει συναδέλφους σε κάθε άλλη νομοθετική επιτροπή που μπορεί να γεφυρώνει ε, τα κενά μεταξύ δικής μας επιτροπής και των άλλων. Γεφυρώνει τις εργασίες μας. Πολύ καλό αυτό. Και πρέπει να αυξήσουμε αυτού του είδους τη συνεργασία. Να ενισχύσουμε στο μέλλον αυτή τη συνεργασία της άλλης επιτροπής. Ο κ. Βοητσετσόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την αναφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Υποστηρίζω πλήρως τις ιδέες που διαπνέουν την αναφορά. Είμαι Πολωνός. Στην Πολωνία το αλογίσιο κρέας δεν καταναλώνεται. Με κάποιες εξαιρέσεις. Για μας ένα άλογο έχει ιδιαίτερη θέση στην παράδοσή μας, στην ιστορία μας δεν έχουμε μεγάλη παράδοση κατανάλωσης αλογίσιου κρέας. Αν εξαρτέταν από μένα, εγώ με τα χαράς θα υποστήριζα την απαγόρευση της καταναλώσεως αλογίσιου κρέατος. Διότι είναι ζώα που είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο, όπως είναι οι γάτες, όπως είναι οι σκύλοι, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους και στάση απέναντί τους. Τέλος πάντων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Πολύ συχνά λοιπόν τα άλογα εκτεύονται για κατανάλωση και δεν νομίζουμε ότι αυτό μπορούμε να τα αλλάξουμε. Το άλογο όμως είναι το μόνο ζώο που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Φερρυπίν. Πολύ συχνά τα άλογα αθλητισμού μετά καταναλώνονται σαν αλογίσιο κρέας στην Ευρώπη. Καμιά φορά πιθανότατα τρώμε εκείνα τα άλογα που είχαν αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να εγγυηθούμε την καλύτερη δυνατή μεταχείριση εκείνων των ζώων που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι δυνατότητες υπάρχουν και που προσφέρονται από κτηνιατρικές διατάξεις θα πρέπει να έχουμε ύψιστες προδιαγραφές όσον αφορά τους ελέγχους, ούτω ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε την ευημερία των ζώων αυτών. Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να υποστηρίξω την αναφορά. Χαίρομαι που υπευλήθη και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρότατα. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους ομιλητές στον κατάλογό μου, λέει Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο ξανά ε, στην αναφέρουσα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θετική ανταπόκριση σε αυτήν την ε, αναφορά. Ένα από αυτά που είπε ο κύριος Βοητσεχόφσκι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι ζώα που χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό και δεν θα έπρεπε να καταλήγουν στη διατροφική αλυσίδα γιατί υπάρχουν ε, αντιφλεγμονώδη, διάφορα φάρμακα ε, τα οποία αν ε, χρησιμοποιούνται σε κάποια άλογα πρέπει αυτά να αποκλείονται από τη διατροφική αλυσίδα. Ξέρουμε όμως ότι τα άλογα του υποδρόμου πολλές φορές ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο ε, τα στέλνουμε εκτός συνόρων, σφαγιάζονται εκεί και μετά εξάγονται και εισάγονται πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν ε, πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα ε, με τους ελέγχους όταν μιλάμε για ε, άλογα για τα οποία δεν υπήρξαν για όλη τη διάρκεια τη ζωή τους στα ιστορικά αρχεία που είναι η περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχουν πάντοτε ιατρικά αρχεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουν στη διατροφική αλυσίδα τα άλογα αυτά γιατί είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του κάθε συνοδευτικού ε, των ζώων αυτών εγγράφου. 70% των ε, αλόγων σφαγιάζονται στον Καναδά. Εμείς είμαστε η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγή για τι χώρε αυτέ και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η απέτηση της εξάμηνης διαμονής στη χώρα σφαγιασμού δεν θα λύσει το πρόβλημα με, το άλογα που έχουν ζήσει 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και που τους έχουν χορηγηθεί κάθε λογής φάρμακα και τελικά καταλήγουν να είναι ζώα που παράγουν κρέας για ανθρώπινη κατανάλωση. Χαίρομαι λοιπόν ε, όλος ιδιαίτερος ε, ότι με το ότι η Επιτροπή σας παίρνει πολύ σοβαρά αυτή την αναφορά και έχετε σκοπό να την προωθήσετε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και τη σχέση με τη Συμφωνία ΣΥΤΑ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να προσπαθήσω να συνοψίσω. Και αν συνάδελφοι διαφωνούν, να πάρετε το λόγο. Λοιπόν, προτείνω το εξή. Για την πρώτη αναφορά 7203 ε, του 2015 να την κλείσουμε. Έχουμε ελεύθερη συμφωνία, συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τον ε, Καναδά, αλλά ε, μπορούμε να τη στείλουμε στην Ίντα και στην ΕΜΒΗ για ενημέρωσή τους και για την άλλη ε, για την άλλη αναφορά ε, έχουμε πολύ περισσότερους ενδιασμούς. Ε, υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας της υγείας. Μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων για το θέμα αυτό γιατί μπορεί να έχουμε στοιχεία τα οποία θα μας χρησιμεύσουν ε, και σε επόμενες αναφορές για το θέμα αυτό. Και τις δύο όμως θα τις προωθήσουμε στην Ίντα και στην Έμβη υπομορφή ε, ε, επιστολής. Θα κλείσουμε λοιπόν τη 0723 και θα αφήσουμε ανοιχτή την 1129 γιατί είναι πολύ ευρύτερο το, το πρίσμα της. Έχουμε όμως και την ε, συμφωνία ΣΥΤΑ με τον Καναδά και έτσι είναι... Ε, έχουμε κάπως, μας έχουν ξεπεράσει εξελίξεις συμφωνείτε ναι Καταρχήν συμφωνώ, αλλά για να είμαστε σαφείς, ε, η συμφωνία συναλλαγών με τον Καναδά έχει ολοκληρωθεί ως προς τη διαπραγματεύση της, αλλά δεν έχει επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο. Ε, αναμένεται να ε, επικυρωθεί, αλλά εντάξει, μπορεί οι διαπραγματεύσεις να μην ξαναρχίσουν, απλώς θέλω να το πω για να είναι σαφές ότι δεν είναι τελειωμένη υπόθεση όσον αφορά, τη όσον αφορά την ε, επικύρωση της συμφωνίας αυτής. Πρόεδρος, το πλαίσιο της αναφοράς αυτής, ε, της σύνταξή της και της υποπολίτης εμάς, ε, είναι διαφορετική Νομίζω ότι το περιεχόμενό της είναι σημαντικό για τις επιτροπές που ανέφερα. Πρέπει να την προωθήσουμε σε αυτές. Και η δεύτερη από τις δύο αναφορές, ε, επειδή δεν είναι μια ε, κατακάθαρη υπόθεση, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Βλέπω ότι όλοι γνέφουν καταφατικά, οπότε πολύ ωραία να προχωρήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την αναφέρουσα που μας διαφώτισε ε, και για τη δική της αναφορά αλλά και για το ευρύτερο θέμα το οποίο πραγματεύεται η αναφορά της και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή. Να περάσουμε τώρα στο 14. Που είναι η αφορά μόνο 812. Oh, who? Who? Mrs. Hasekamp, please. παρακαλώ κύριε Hasekamp, δεν σας είδα. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Could you use the microphone, please? Um, ναι, συγγνώμη. Συμφωνώ με το συμπέρασμά σας, αλλά θέλω... Ε, ρώτησα κάποια πράγματα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να μου απαντήσουν. Για να ρίξει λίγο φως στην υπόθεση ή αργότερα. Έχουμε ε, αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ δεδομένο ότι θα σας απαντήσουν. Σε ερωτήσεις της κυρίας Χάζεκαμπ μπορείτε γραπτός να απευθύνετε στη γραμματεία. Σύντομες απαντήσεις, έτσι, ας προχωρήσουμε. Ε, λοιπόν, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την κυρία Χάζεκαμπ που υπογράμμισε αυτή την υπόθεση. Ωραία, τώρα θα πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το υπαριθμό 14 σημείων αναφορά 8-12. Αποουσιάζει αναφέρον, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Στέφαν Φάντερ Σπίγκελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πόσο εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συνεισφορά των αιμοδοτών στα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Είναι πολύτιμο. Καμία χειρουργική, καμία ε, αιματολογία, ογκολογία, ε, αντιμετώπιση τραυμάτων δεν θα μπορούσε να ε, διανοηθεί κανείς χωρίς αιμοδοσία των πολιτών. Έχει σημασία όμως να καταλάβουμε ότι για να καταλήξουμε και να φτάσουμε σε αυτές τις θεραπείες ε, χρειάζεται ε, μία ολόκληρη αλυσίδα και περίπλοκη ε, διαδικασιών, όπως λέει και ο αναφέρον. Κάποια πρώτα βήματα είναι τα βήματα του αιμοδότη, που είναι η συλλογή του αίματος, η αιμοληψία δηλαδή, ο έλεγχος κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δύο οι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει το πλάσμα του αίματος. Το πρώτο, όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, είναι να στέλνονται σε νοσοκομεία όπως χρησιμοποιούνται για διάφορα προβλήματα αιμορραγίας ε, κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου και αυτή είναι η κλασική ε, δουλειά κάποιων κρατικών ή μη κρατικών φορέων όπως είναι ο Ερυθρός Σταυρός γιατί είναι και μόνιμη η ζήτηση. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει το πλάσμα του αίματος είναι να σταλεί σε ε, εταιρείε που παράγουν φαρμακευτικά προϊόντα και υπάρχει μια ολόκληρη ε, διαδικασία διήθησης για τα παράγωγα πλάσματος που είναι ε, προϊόντα που έχουν να κάνουν με την αιμοσφαιρίνη ή για αιμοφιλικούς και άλλους που έχουν προβλήματα ανοσοποιητικού. Αυτά τα αναλαμβάνουν ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες και είναι ένας κλάδος με αυξανόμενη ζήτηση. Γι' αυτό υπάρχει και κοινοτική νομοθεσία ευρωπαϊκή, ε, που διπλή, δηλαδή δεν ε, είναι ίδια. Το πρώτο με τους αιμοδότες ε, και την αιμοληψία έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αίματος για το πώς διανέμονται αυτά και στα νοσοκομεία για μεταγγίσεις. Όμως όταν πρόκειται για το πλάσμα το οποίο το στέλνουν σε φαρμακευτικές εταιρείες, ιδιωτικέ επαναλαμβάνω, για την παραγωγή, τότε ε, ε, εκεί επεμβαίνει και ισχύει η νομοθεσία για τα φάρμακα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζει το πεδίο εφαρμογή αυτών των νομοθετημάτων, είτε η νομοθεσία για το αίμα είτε για τα φάρμακα μόνο σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Όταν μιλούμε για θέματα οικονομικά ή βιοηθικά, όπως λέει η αναφορά, αυτά εμπίπτουν εντελώς στην εθνική νομοθεσία των 28 κρατών μελών. Τώρα, σε περίπτωση που είναι αμοιβόμενη αιμοδοσία, γιατί αυτό λέει ο αναφέρον ότι εκεί μπαίνουν ηθικά ζητήματα, ενώ κανονικά για μας η ομοδοσία θα πρέπει να είναι εθελοντική και μη αμοιβόμενη. Ε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι επαγγελματίε της υγείας θεωρούν ότι Όταν ε, πληρώνεις για ε, έναν αιμοδότη μπορεί εκείνος ακριβώς επειδή έχει το οικονομικό κίνητρο να αποκρύψει στοιχεία που είναι κρίσιμα για την ποιότητα και την ασφάλεια. Ενώ όταν είναι θελοντική η νομοθεσία, ε, συγγνώμη, η αιμοδοσία υπάρχει μικρότερος κίνδυνος. Οπότε η ίδια η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το αίμα και για τα φάρμακα ζητεί να ενθαρρύνονται έντονα, να παροτρύνονται τα κράτη-μέλη ότι θα παραμένει η αιμοδοσία εθελοντική και μη αμοιβόμενη. Αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά όταν θέλουν τα κράτη-μέλη μπορούν να το κάνουν σε εθνικό επίπεδο, δια νόμου, υποχρεωτικό. Και ξέρουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη απαγορεύεται η αμοιβή. Και αυτό αντανακλά την πραγματικότητα στον κλάδο αυτό. Πολλά είναι εκείνα τα κράτη-μέλη που απαιτούν ε, δωρεάν εθελοντική αιμοδοσία και υπάρχουν και κάποια άλλα όπου η δραστηριότητα αιμοληψίας, η λήψης πλάσματος για φαρμακευτικά ε, μέσα είναι σημαντικά και για την ε, παροχή και για τη ζήτηση και για την προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε μία έκθεση που πρόκειται να, εκδώσει, να δημοσιεύσει προσεχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την νομοθεσία περί ε, αίματος και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εθελοντική και μη αμοιβόμενη αιμοδοσία. Τα περισσότερα κράτη-μέλη ζητούν να εφαρμοστεί αυτή η αρχή, ωστόσο στην πράξη η εφαρμογή χωλαίνει δεν είναι ούτε τόσο εύκολη και μάλιστα διαφέρει και ποικίλει από χώρα σε χώρα. Δεν είναι εύκολο να γίνει καλή διάκριση ανάμεσα στο στο στο συνιστά πληρωμή, αμοιβή ή ανταμοιβή, αποζημίωση. Α πούμε, άλλο είναι να πληρώσει ένα αιμοδότη για να δώσει αίμα και άλλο είναι να του πληρώσει, να του αποζημιώσει το εισιτήριο του λεωφορείου που θα πάει στο κέντρο αιμοδοσία για να δώσει αίμα. Σε πολλά κράτη-μέλη διαφέρει η κατάσταση λοιπόν. Δεν είναι τόσο σαφή και ξεκάθαρα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο συνάδελφο θέλει το λόγο. κυρία Βεθέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ε, εξαντλητική απάντηση και σε λεπτομέρειες και που μας είπατε ότι αυτή η συγκριτική έκθεση για το πώς εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα κράτη-μέλη θα ε, δημοσιευθεί προσεχώς. Προσεχώς πότε, εντός του 15, εντός του μηνός, όπως προβλεπόταν, θα μου απαντήσετε στη συνέχεια. Αυτό που ήθελα να τονίσω κυρίως είναι ότι πέρα από τις αρχές της επικουρικότητας που φυσικά ε, ε, βρίσκουν το εφαρμογή και τα βιοειθικά και τα διαντολογικά ζητήματα, τα φάρμακα που είναι παράγωγα πλάσματος, ανθρωπίνου αίματος, χρησιμοποιούνται και περισσότερο. Χρησιμεύουν για πολλές ασθένειες και η βιομηχανία τα προτιμάει και έχουν και αυτό το πλαίσιο ότι δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, για τα φάρμακα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που καλύπτονται από ρυθμίσεις εδώ και 12-13 χρόνια, έτσι δεν είναι και από την ενημέρωση που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να μου απαντήσετε ε, πώς το βλέπετε και πώς το περιμένετε. Δεν αναμένεται αναθεώρηση αυτής της νομοθεσίας όταν το γενικότερο πλαίσιο για τα φάρμακα ε, αναθεωρείται. Εδώ στο Κοινοβούλιο μας απασχολεί αυτό και στην κοινωνία των πολιτών παντού το σημερινό ε, μοντέλο πρόσβαση στα φάρμακα που έχει να κάνει με διπλώματα έβριση τεχνίας, με παραγωγή φαρμάκων και με δημόσιες επενδύσεις ε, στην ε, φαρμακευτική έρευνα και παραγωγή και παρασκευή φαρμάκων χρειάζεται κάποια προσαρμογή. Άρα λοιπόν από τη δική μας επιτροπή θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς πρώτον. Να, διότι ο συνάδελφος προηγουμένως. Για το προηγούμενο θέμα, για το κρέας του αλόγου, να ε, το διαβιβάσουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ΕΝΒΗ που έχει και τις δυνατότητες και τις γνώσεις να μας πει τι πρέπει να κάνουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει παρακαλώ εάν έχει καμιά ιδέα ή αν σκέφτεται ότι κάπως πρέπει να ε, πλαισιώσει την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας ή αυτών των οδηγιών στο πώς έχει πρόσβαση στα φάρμακα, η έρευνα κτλ. Εμεί να ζητήσουμε και από τον ΕΟΦ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τη γνώμη του, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η θέση και η άποψή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. I have no... Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, αλλά θα ήθελα να κάνω εγώ μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε άλλωστε και η κυρία Μπεσέρα, η αναφορά στην έρευνα που έχει κάνει σε επίπεδο κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί και των μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών για την ενθάρρυνση της εθελοντικής και μη αμοιβόμενη ε, αιμοδοσίας. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει μία έκθεση η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί μέχρι το τέλος του έτους. Το έτος όμως τελειώνει. Πότε θα το δούμε, πότε θα τη δούμε αυτή την ε, έκθεση. Παρακαλώ απαντήστε μας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Η έκθεση, να σας πω με κάθε ειλικρίνεια, θα είναι για τις αρχές του 2016. Πραγματικά όμως σε εσωτερικό επίπεδο είμαστε στο τελικό στάδιο ολοκληρώνουμε αυτήν την έκθεση εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σύντομα λοιπόν θα λάβετε γνώση αυτής της έκθεσης που ε, πραγματεύεται ακριβώς πώς ε, αντιμετωπίζουν το θέμα της εθελοντικής και μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας ε, τα κράτη-μέλη αλλά και το ευρύτερο θέμα της νομοθεσίας περί αίματος, πώς δηλαδή οι διάφορες απαιτήσει εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη και όπως είπατε και εσείς, η νομοθεσία αυτή τη στιγμή είναι 12 ετών ήδη. Δεν θα πω αν χρειάζεται αναθεώρηση ή όχι, αλλά τουλάχιστον όταν θα δημοσιευθεί αυτή η έκθεση θα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Οι συνάδελφοι δεν έχουν προτείνει τίποτε. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ. Εγώ λοιπόν έχω το δύσκολο καθήκον να συνοψίσω κατά τη γνώμη μου, να την κρατήσουμε ανοιχτή μέχρι την τελική έκθεση και όταν δημοσιευτεί η έκθεση ευχαρίστω να τη διαβάσω και να προωθήσουμε την αναφορά μαζί με την έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όπως είπε και η κυρία Μπεθέρα. Και ίσως να μείνουμε και σε επαφή με τον ε, Οργανισμό Φαρμάκων μήπως έχουν επιπλέον πληροφορίες. Εμείς συνεργαζόμαστε πολύ εργαζόμαστε με, την, ε, τον Οργανισμό Φαρμάκων τον Ευρωπαϊκό, πολύ στενά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε μας γλιτώνεται και από τον κόπο και την προσπάθεια. Το εκτιμούμε, λέει η εν πάση περιπτώσει. Ίσως δεν ήμουν ξεκάθαρο στην εξήγησή μου. Ακόμα κι αν εκείνα τα προϊόντα εμπίπτουν στον τομέα νομοθεσίας περί φαρμακευτικών προϊόντων, λοιπόν μιλάμε εδώ για την εθελοντική ή μη αιμοδοσία. Αυτά τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, ε, θα εμπέσουν στην νομοθεσία περί αίματος. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους, τους υπευθύνους για τα φαρμακευτικά, διότι ξέρουμε ότι μια αλλαγή των κριτηρίων αφορά τον τομέα αυτό ίσως επηρεάσει και τα φάρμακα. Οπότε υπάρχει μια στενή διασύνδεση. Πολύ ενδιαφέρον τομέας λέει η Πρόεδρος και προσβλέπουμε στη δημοσίευση της εκθέσεως και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρότεινα. Παραμένει ανοιχτή, περιμένουμε για τη δημοσίευση της εκθέσεως θα τη διαβάσουμε, θα τη χωνέψουμε και θα στείλουμε αυτή την αναφορά προς ενημέρωση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Καλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας προχωρήσουμε και πάμε στο σημείο 15. Είναι η αναφορά 43 του 2014 για τη γενική απαγόρευση της κυκλοφενάκης. Είναι μοναδική περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται από έναν Ευρωβουλευτή, την Μπεατρίς Πεσέρα. Η αναφέρουσα, αναφέρον, εκπροσωπείται. Ευχαριστώ, ναι. Εκπροσωπώ εδώ και μιλώ εξ ονόματος ε, ενός αναφέροντος για μια αυτή τη ε, αναφορά. Είναι κάπως περίεργο από την αρχή αυτό. Γιατί μιλήσαμε για τα παιδιά, μετά μπήκαμε σε θέματα φαρμακευτικά και διατροφικής ασφάλειας και τώρα ε, θα μιλήσουμε για ε, περιβάλλον, για ε, εξοικονόμηση ενέργειας και για μια σειρά θέματα που έχουν να κάνουν με το Κοινοβούλιο γενικά όλα τα θέματα είναι εγκάρσια. Εδώ είναι ένα φάρμακο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε σε διάφορα κράτη-μέλη στην Ισπανία το 2013 και η Ευρωπαϊκή, Οργανισμός ε, Φαρμάκων σε μία έκθεση ε, στα ε, χειροειδή και στις αγελάδες το απογόρευσε. Γιατί μιλάμε για τη σημασία να τι σημασία έχει η δικλοφενάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχει ε, ε, ε, πάνω από 90% των ζώων των, των αρπακτικών, των ορνέων και οι γήπες από διάφορα είδη τρώνε πολλά πτώματα ζώων ε, και βοηθούν ε, στην ε, αποφυγή σύψης αυτών των πτωμάτων και μόλυσης του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία αυτή, ο οργανισμός, δεν λέει ότι πρέπει να απογορευτεί τελείως η χρήση ε, στα ζώα, αλλά πρέπει να περιοριστεί και να υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης για να μην κινδυνεύσουν ε, τα ζώα αυτά τα αρπακτικά γήπες. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν εγώ ότι υπάρχει ένα σημείο που είναι σαφής η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ζημιά στο περιβάλλον, που μολύνεται έτσι κι αλλιώς, γιατί σας είπα ότι έχουμε τόσο μεγάλο πληθυσμό, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προστατεύουν τα άγρια πτηνά όπως ορίζει η Οδηγία 147 του 2009 και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά της δικλοφενάκης και αλλού όπως ε, στην ε, Σύνοδο Κορυφής για την Άγρια Πανίδα του ΟΗΕ για να απαγορευτεί αυτό το φάρμακο γιατί είναι επικίνδυνο για την Άγρια Πανίδα. Μια που έχω το λόγο εδώ θέλετε να σας πω και τη δική μου άποψη. Αυτά τα λέω εξ ονόματος του αναφέροντος. Αλλά και προσωπικά θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Τι προτείνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη την ειδική κατάσταση της Ισπανίας και να ζητήσουν ειδική απάντηση από την Ισπανική ε, κυβέρνηση για την προστασία των γηπών και λοιπόν αρπακτικών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει με τα μέτρα που πρότεινε ο ΕΟΦ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, υπάρχει καμιά εποπτεία, καμιά παρακολούθηση για το εθνικό σχέδιο. Έχουν ε, παρατηρηθεί ε, οι επιπτώσεις ε, στην άγρια πανίδα στις χώρες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτού του φαρμάκου και ποια είναι η δυνατότητα να καταφύγουμε σε ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις και αυλαβής. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η κτηνοτροφία. Είναι πολύ σημαντικό, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυκλική οικονομία. Και αυτό κυκλική οικονομία είναι, ανακύκλωση κάνουν τα όρνεα για το περιβάλλον και είναι και πλούτος και ε, θέμα δημόσιας υγείας. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην ανάπτυξη και τι μαθήματα μπορούμε να ε, ε, έχουμε και διδάγματα να εξάγουμε από τα όσα ε, έγιναν στην Ινδία και στην Ασία και τι σήμαινε αυτό για τα άγρια ζώα που τρέφονται με πτώματα ζώων, νεκροφάγα. And Και τώρα Θέλουμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτό. Αριάν Βαντεστάπεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή. Η κυρία Βουλευτή Συνόψη άριστα την παρούσα κατάσταση, διότι αναφορά κατετέθη Φεβρουάριο 2014. Οπότε σήμερα είμαστε τέλος 2015 και τα λάβαμε αυτά υπόψη να επενθυμίσω κάτι. Κατανοούμε αυτή όταν επετράπη η κυκλοφορία της στην Ισπανία, επετράπη, δημιούργησε ανησυχία. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια όρνεα. Από το 1993 είναι αυτή η ουσία στην ευρωπαϊκή αγορά και καμία περίπτωση δηλητηρίασης των ορνέων δεν διαπιστώθηκε μέχρι τώρα. Είναι κάτι σημαντικό δεν είναι κάτι καινούριο όσον αφορά τη χρήση του φαρμάκου αυτού. Βεβαίως εξετάσαμε όλες τις διεξόδους, όλες τις λύσεις και η απαγόρευση ή μάλλον η απόσυρση της αδειοδότησης του φαρμάκου αυτού είναι κάτι που ζητήθηκε από κάποιους αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα στοιχείο συγκεκριμένο που μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να ξέρετε ότι η νομοθεσία περί φαρμάκων ε, είτε για τους ανθρώπους είτε κτηνιατρικά αφορά τις σχέσεις, ε, εξετάζεται βάση της σχέσης κόστους αφέλους και σύμφωνα με την γνωμοδότηση που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αυτό το ποσοστό ωφέλους κινδύνου παραμένει θετικό. Άρα δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε. Επιπλέον όπως σωστά αναφέρατε πρόκειται περί φαρμάκου είναι κτηνιατρικά φάρμακα που αντιδοτούνται σε εθνικό επίπεδο σε πέντε σήμερα. Εξάλλου φαίνεται ότι η κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά το, τη δικλοφενάκη και τα όρνια είναι διαφορετικά. Σε κάποια κάτι μέλη δεν επιτρέπεται αυτό το φάρμακο να κυκλοφορεί στη χώρα και δεν έχουν κανένα πληθυσμό ορνέων. Για να τα γνωρίζετε λοιπόν. Μόνο δύο κράτη-μέλη θα εξέταζαν το ενδεχόμενο αποσύρσεω τη αδειοδοτήσεω. Αυτά τα δύο κράτη-μέλη δεν έχουν ούτε όρνια ούτε ποτέ είχαν επιτρέψει την δικλοφενάκη. Είναι πολύ ε, ιδιαίτερη κατάσταση. Για να παραδείγουμε τώρα στα κάτι μέλη τα οποία έχουν το φάρμακο, το έχουν αδειοδοτήσει σε εθνικό επίπεδο και έχουν πληθυσμό ορνέων, ένα σχέδιο δράσεως ζητήθηκε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάσε δύο φορές μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ήρθε σε επαφή με τα κράτη-μέλη ούτως ώστε ε, να μπορέσουν να μα δώσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεως δηλαδή τι μέτρα θέλουν να κάνουν για να μειώσουν τον κίνδυνο ή έχουν δρομολογήσει ή θέλουν να δρομολογήσουν μέσω γραπτής ενημέρωσης. Λοιπόν, θα πρέπει να συμπεραβάνετε στο έγγραφο των μετρών που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη. Είναι δημοσιευμένα στην σελίδα μας τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη. Ε, πριν από μερικούς μήνες δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο. Έκτοτε δεν έχουμε ε, κάποια αντίδραση από την κοινωνία των πολιτών ή εκείνους που είχαν κάνει σχόλια όσον αφορά αυτό το σημαντικό ζήτημα. Αυτό που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες είναι βάση της πραγματικής εφαρμογής των σχεδίων δράσεως θα κρίνουμε. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ένοχο ένα κράτος μέλος όταν δεν έχει ένα καλό σχέδιο κράτος χωρίς, χωρίς στοιχεία. Η Ισπανία είναι ένα από τα άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι σαφή ε, η ικανότητα να αντιμετωπίσουν το κίνδυνο μέσω των σχεδίων ε, χειρισμού ε, του κινδύνου και του σχεδίου δράσεως. Υπάρχει κίνδυνος αν χρησιμοποιούμε τη δικλοφενάκη σε κάποια ζώα, αν εγκαταλείπονται στα λιβάδια αυτά τα ζώα και δεν έχουν εφαρμοστεί τα βέοντα. Θεωρείται ελάχιστο ο κίνδυνος που δημιουργείται όμως και μπορεί να συγκρατηθεί και να ελεγχθεί αν τα μέτρα, τα σχετικά για τη συγκράτηση του κινδύνου είναι αποτελεσματικά. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε αρχές ε, του 2016 από, την, ε, από όταν θα έχουμε κάποιες μήνες εμπειρίες από τα σχέδια δράσης είναι να δούμε τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη σαν τα σχέδια δράσης, δηλαδή τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, τα αποτελέσματα των ενσημένων ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις, εκεί που υπάρχει ε, εντατική κτηνοτροφία και να δούμε τα αποτελέσματα. Εάν στα, επίσης, στα επίπεδα μονίμων επιτροπών δεν αρκούν. Μπορούμε να αποστείλουμε και κτηνιάτρους της Διευθύνσεως Αρμοδίας που ασχολείται με τους ελέγχους στα κράτη-μέλη και να δούμε πώς εφαρμόζονται τα σχέδια δράσης στην πραγματικότητα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είστε βέβαιοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για μας. Ότι το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε θα ήταν να δημιουργηθεί μια κατάσταση κατά την οποία ακόμα και πολύ ε, λιγότερα συμβούν από αυτά που συνέβησαν στην ε, Ινδική υποήπειρο. Λοιπόν, με την νομοθεσία που έχουμε για τα φάρμακα, είναι το καλύτερα μέτρα αυτά που λάβαμε, που θα μπορούσαμε να λάβουμε. Υπάρχει και ένα άλλο φάρμακο που θα μπορούσαμε ότι είναι κάπω παρόμοιο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ενθαρρυνεί τη χρήση ενό φαρμάκου έναντι άλλου. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε ένα φάρμακο βάσει του γεγονότο ότι δεν υπάρχει άλλο, μέχρι να αποδείξει τον εναντίου. Αν αποδειχθεί ότι το φάρμακο μπορεί να δημιουργήσει ε, πρόβλημα στους πληθυσμούς των Ορνέων. Μέχρι τώρα και ευτυχώ όμως δεν έχουμε καμία τέτοια σχετική ενημέρωση, απόδειξη περί προβλημάτων στην Ευρώπη που δημιουργούνται στην Ευρώπη λόγω αυτού του φαρμάκου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε. Μπορεί να μιλήσουν συνάδελφοι. Δεν είναι πολύ στην αίθουσα. Πέμπτη απόγευμα βλέπετε και φεύγουν οι πτήσεις, επιστρέφουν στις χώρες τους. Δυστυχώ αυτό ισχύει και για μένα. Πρέπει να περιμένω μέχρι την Παρασκευή να γυρίσω στην πατρίδα μου, στο σπίτι μου. Ελπίζω αυτό να αλλάξει του χρόνου. Τώρα λοιπόν κάνει δεν ζήτησε το λόγο, οπότε να δώσω το λόγο ξανά στην αναφέρουσα για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο εξαντλητική ε, εξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και την τόσο στεναρή. Θέλω να πω το εξής κινδυνεύει με εξαφάνιση αυτό, το είδος αυτός ο γήπας. Ε, στο περιβάλλον ξέρουμε τι γίνεται και τι σημαίνει για την υγεία. Είδαμε τι έγινε στην ε, ε, Ινδική Υποήπειρο. Στην Ισπανία εγώ πιστεύω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα μας δώσουν στοιχεία και προσβλέπω σε αυτό για το πρόγραμμα δράσης, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ε, λειτουργικότητας ε, γιατί έχουμε τώρα διαδοχικές εκλογές στην Ισπανία. Εδώ και ένα χρόνο είχαμε διαδοχικές εκλογές και τώρα έχουμε βουλευτικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι μήνες ολόκληρος είμαστε σε παράλυση και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένη δράση παραμονές εκλογών τώρα και πόσο μάλλον για τέτοια θέματα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αυτό που θα γίνει μέσα σε δύο μήνες είναι σημαντικό γιατί η ζημιά δεν επανορθώνεται οπότε θα ήθελα παρακαλώ στο μεταξύ να αναλυφθεί κάποια δράση και να γνωρίζει η Ισπανική κυβέρνηση ότι και το παρακολουθούμε, αλλά θέλουμε να δούμε επιχειρησιακά τι θα κάνουν. Και με τον Ισπανικό Οργανισμό Φαρμάκων, τι μέτρα προβλέπουν και πόσο ασφαλής είναι η χρήση αυτού του φαρμάκου δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσουν μήνες, δεν είναι ανώδυνο το θέμα. Να έχουμε άιντε τράτο μεγάλο, χρονικό. Και ο, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ζητήσει ρητά την απόσυρση του φαρμάκου όταν βλέπουμε τέτοιες ζημίες. Τώρα λέτε δεν έχουμε εγγυήσει ότι γίνονται. Εντάξει. Θα πρέπει και η δική μας επιτροπή να το παρακολουθήσει το θέμα. Για ε, αυτή τη στιγμή λάβουμε την απάντηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Uh, Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σαφώς παρουσίασε την κατάσταση. Όμως θα θέλαμε ο αναφέρον ε, να μας δώσει περισσότερα ε, στοιχεία. Πρέπει να έχουμε επαρκέστερα στοιχεία. Προτείνω το εξής να βάλουμε μια προθεσμία δύο μήνες από τώρα. Και σε αυτή την περίοδο δύο μηνών μπορεί ο αναφέρον να αποστείλει στη γραμματεία ε, περισσότερες ε, πληροφορίες για να στηρίξει αυτήν την αναφορά. Συμφωνείτε? Βεβαίω τα στοιχεία αυτά θα τα προωθήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ λοιπόν ε, στείλετε τα επιπλέον στοιχεία στην ε, γραμματεία μας. Θα ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως την αφήνουμε ε, ανοιχτή αναμένοντας τις πληροφορίες από τον αναφέροντα. Ωραία. Φτάνουμε σιγά σιγά στο επόμενο σημείο την αναφορά 59 του 2011 Φολφχαντ Μπέμπερ γερμανικής ηθαγένεια, ε, για εικαζόμενη παραβίαση οδηγίας ε, ε, κτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με την άδεια λειτουργίας λατομείου λίθου κοντά στο Αλικάντε στην Ισπανία. Δεν είναι εδώ αναφέρον, όμως υπάρχει μια παρουσίαση σε διαφάνειες, ένας slideshow και θα αρχίσουμε με αυτήν. I can I think we can speed up the show a bit. Να το πάμε λίγο πιο γρήγορα ίσως. Η Νατάλια φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Πάμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Λοιπόν, τρεις, αναφορές, τρεις αναφέροντες υπήρχαν στην αρχή. Ένας μόνο επεβίωσε. Ζει πάρα πολύ κοντά σε ένα λατομείο λίθου. Υπάρχουν συνεχώς ε, ανατινάξεις και φαίνεται εκρήξεις, ε, οι οποίες ε, τις οποίες ε, και ένα σεισμογράφος αποδεικνύει. Έχουμε εδώ ένα σεισμογράφημα το οποίο έχει ληφθεί κοντά στο σπίτι του αναφέροντος. Το λατομείο έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του χωρίς, χωρίς άδεια και χωρίς καμία διαβούλευση γιατί η εκτίμαση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έγινε. Αυτά πολύ σύντομα και κάποια στοιχεία για το ιστορικό της υπόθεσης. Είχε υποσχεθεί το Μάρτιο να κλείσει το λατομείο λίθου γιατί υπήρχαν πολλές τέτοιες υποσχέσεις και αποδικαστικές αποφάσεις. Είναι Δεκέμβρη, συνεχίζονται οι δραστηριότητες του λατομείου, αρχίζουν εκρήξεις και σκάψιμο Δευτέρα με Παρασκευή, 6 ώρα το πρωί και ο αναφέρον έχει πραγματικά απειβδίσει, προσπαθεί να πιέσει και να ζητήσει και από άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και την ε, ε, αυτοδιοίκηση της Βαλένθια να κλείσει το λατομείο, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα μετά από τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Πάρα πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό ήταν αυτό το slideshow. Είναι εδώ ο Χωσέ Ράμος, Φλωρίδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, όντως ε, φάνηκε σε αυτά τα slides που έστειλε ο αναφέρον, η αναφορά αυτή έχει σαν αντικείμενο τις εξορρυκτικές δραστηριότητε σε ένα λατομείο ε, στο Δήμο Πέγο που είναι δίπλα στην Αρσούμπια, στην επαρχία Αλικάντε, στην αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθιας στην Ισπανία. Ο αναφέρον στην αναφορά του καταγγέλει ότι το λατομείο αυτό έχει διευρυνθεί το έτος 2007 χωρίς να έχει γίνει καμία μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, χωρίς να υπάρξει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ούτε αξιολόγησης των ε, αποτελεσμάτων και του αντικτύπου αυτής της δραστηριότητα στο περιβάλλον. Ο αναφέρον καταγγέλει όχι απλώς τις ζημιές για το περιβάλλον, αλλά και τον κίνδυνο που σημαίνει για τους περιοίκους η εξορρυκτική αυτή δραστηριότητα στο λόγο λατομείο. Επίσης τονίζει την ε, ε, απραξία των αρμοδίων τοπικών και περιφερειακών αρχών. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επέμβει μόνο σε θέματα που καλύπτονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πρόκειται για το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ένωσης. Έχουμε πει και σε γραπτές προηγούμενες επικοινωνίες μαζί σας και στην τελευταία επιστολή, το Φεβρουάριο φέτος, όπου προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε ε, όλη αυτή την περίπλοκη περίπτωση που και αυτή έχει τραβήξει χρόνια. Τι λέει η περιβαλλοντική νομοθεσία που βρίσκεται εδώ εφαρμογή είναι η οδηγία για τη μελέτη ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου. Επίσης, προστασία της φύσης σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι αυτό το λατομείο έχει ε, επιπτώσεις στην ε, Natura 2000, γιατί και κοντά υπάρχει ένας βιόπιτοπος. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μελέτη αντικτύπου, αναφέρεται στο παράρτημα 1 της οδηγίας ε, και τέτοιου είδους δραστηριότητες, εξορίξει σε μεγάλα λατομεία και στο παράρτημα 2 αναφέρονται άλλου είδους λατομεία και εδώ θα πρέπει οι Ισπανικές αρχές τουλάχιστον να ελέγξουν ε, τις οριακές τιμές ε, της Ισπανικής νομοθεσίας στη μεταφορά της οδηγίας. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω, όπως σας είπα και στη γραπτή μας απάντηση, το λατομείο αυτό λειτουργεί από τη δεκαετία του 40 του περασμένου αιώνα, όταν βεβαίω δεν υπήρχαν νόμοι για προστασία περιβάλλοντος και τα λοιπά όπως υπάρχουν σήμερα. Ούτε ήταν καν μέλος η Ισπανία, ούτε υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τίποτα. Όμως, επειδή αυτή η δραστηριότητα διευρύνθηκε σημαντικά το έτος 2007, αυτό θα απαιτούσε το νέο έργο διεύρυνσης να έχει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έπραξε. Με βάση αυτή την αναφορά και κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου άνοιξε έρευνα με ένα πιλωτικό πρόγραμμα και είχε ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ισπανικές Αρχές όλα αυτά τα χρόνια. Μας ενημέρωσαν τέσσερις φορές οι Ισπανικές Αρχές και αρμόδιες αρχές είναι η αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθια, η περιφερειακή κυβέρνηση δηλαδή, αλλά και η Δήμη Πέγο και Αψούδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν διευκρίνιζε προς τις ισπανικές αρχές ότι θεωρεί ότι εδώ έπρεπε να γίνει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, οπωσδήποτε. Πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την εξέταση αυτού του θέματος διαπιστώσαμε ότι επενέβησαν οι εθνικές αρχές. Ε, ο ντόπιο συνήγορος του πολίτη ε, ξεκίνησε έρευνα και ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αυτής της εμπορικής δραστηριότητας. Και όπως προηγουμένως υπόθηκε υπάρχουν και διάφοροι σύλλογοι και οργανώσεις ε, που ε, προσέφηγαν κατά της ολιγορίας ή της αδράνειας των αρχών και υπάρχουν και διάφορες δικαστικές αποφάσεις. Η μία από το Φεβρουάριο του 2013 από Διοικητικό Δικαστήριο του Αλικάντε και στη συνέχεια απόφαση ε, του ε, Ανώτερου Δικαστηρίου στη Βαλένθια του Σεπτέμβριο 2014. Έχει τώρα τα στοιχεία στη γραπτή απάντησή μας, όπου ε, ουσιαστικά τι λένε, ότι αυτή η δραστηριότητα δεν έχει άδεια ούτε για, το περιβάλλον, ούτε καν για τη λειτουργία της. Και θα πρέπει να σταματήσει, ε, να πάυσει η δραστηριότητα αυτή. Και αν θέλουν να ξαναρχίσουν την εξόριξη, δηλαδή τη λειτουργία του νταμαριού, θα πρέπει να ζητήσουν ε, τις απαραίτητες άδειε από τη διοίκηση, Καινούρια άδεια δηλαδή. Και προηγουμένως να γίνει περιβαλλοντική μελέτη του έργου. Έκτοτε λοιπόν τι έχει συμβεί. Η λόγω επιχείρηση είχε, όπως είχε δικαίωμα, έχει προσφύγει. Γιατί είναι κράτο δικαίου και κοινότητα δικαίου. Έκανε προσφυγή, έφεσε δηλαδή σε αυτή την απόφαση των δικαστηρίων που ακόμα εκκρεμούν στη δικαιοσύνη τα ζητήματα και οι αρμόδιες διοικητικέ αρχές, δηλαδή και οι Δήμοι, αλλά και η Γενεραλίτα Τουαλετσιάνα, που είναι η περιφερειακή κυβέρνηση και έχει τι βασικέ αρμοδιότητες στο θέμα αυτό, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και ζητούν τη διακοπή λειτουργίας του λατομείου. Κάνουν και επιθεωρήσεις. Και ζητήθηκε από την επιχείρηση να σταματήσει τη δράση, όπως ε, ανέφερα προηγουμένως. Να σταματήσει η λειτουργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως ως θεματοφύλακας των συνθήκων θα μπορούσε να αρχίσει ε, να προσφύγει στο δικαστήριο επί παραλήψη κατά του Βασιλείου της Ισπανίας για μη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Αλλά οι αρμόδιες ισπανικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν προς το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εμπλέκονται και εθνικά δικαστήρια και ο εθνικός δικαστής είναι και κοινοτικός δικαστής κατεξοχήν. Το μόνο που θα μπορούσαμε να πετύχουμε μετά από πολλά χρόνια είναι να αποφανθεί το ε, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά στο μεταξύ δεν θα μπορούσαν τα εθνικά δικαστήρια να επιβάλλουν ούτε την πάυση της λειτουργίας, ούτε την αποζημίωση των περιοίκων, όπως γίνεται με την εθνική δικαιοδοσία. Έχουμε απευθυνθεί και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν οι περίοικοι που έχουν υποστεί βλάβη και ζημία να ζητήσουν αποζημίωση από αυτή την παράνομη δραστηριότητα και τη λαθρέα λειτουργία του λατομείου. Οπότε είναι πολύ πιο αποτελεσματική η δράση των εθνικών δικαστηρίων και δεν ε, χρειάζεται να προσφύγουμε. Και οι περίοικοι λοιπόν και οι συλλογοί θα πρέπει να απαιτήσουν την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Αυτό δεν έχει ζητηθεί εξ όσων γνωρίζουμε Υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων να σταματήσει η λειτουργία, δηλαδή μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, γιατί εκκρεμεί η έφεση. Και σε σχέση με τα όσα σας είπαμε την περασμένη φορά, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, οπότε δεν έχει νόημα να επέμβει η Κομισιόν. Ακόμα όμως και αν ισχύει αυτό, ε, είπαμε στις Ισπανικές Αρχές ότι θέλουμε να παρακολουθήσουμε την έκβαση και πριν από ένα μήνα λάβαμε την πληροφόρηση και από τους δύο Δήμους ε, που θίγονται και από την περιφερειακή κυβέρνηση και μας είπαν ότι έχει κάνει έφεση η εταιρεία και ξέρω ότι ο αναφέρον λέει ότι συνεχίζονται οι εκρήξεις και οι ε, εξορίξεις, αλλά η τελευταία έκρηξη ήταν τον Ιούνιο φέτος ε, και έκτοτε δεν έχει εγκριθεί καμία τέτοια δραστηριότητα. Και επίσημα ενημερώθηκε η εταιρεία ότι θα πρέπει να αναστείλει απολύτω τη λειτουργία της μέχρι να εκδοθούν οι τελικές δικαστικές αποφάσεις. Και αν θέλει να συνεχίσει η δραστηριότητα πρέπει να καταθέσει ένα νέο σχέδιο και να περιμένει να γίνει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Συνοψίζω. Έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρέμβει. Ανησύχησε από την αδράνεια των αρχών. Ευχαριστούμε τους αναφέροντες που έθεσαν υπόψη μας στη συγκεκριμένη περίπτωση κακής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτεραιότητες, τη μη συμμόρφωση, τη μη μεταφορά των οδηγιών, ενώ αυτή τη φορά δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά ε, είναι ένα ζήτημα εθνικών δικαστηρίων. Και φτάνει αυτό για να εφαρμοστεί σωστά και να επιβληθεί η εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, θέλετε να πάρετε το λόγο. Jude. Ευχαριστώ πολύ. Το γεγονός ε, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτέ εδώ, να πω κι εγώ ότι είναι πραγματικά μάλλον άσχημο να μένει κανεί δίπλα σε ένα λατομείο λίθου που ε, δηλητηριάζει τη ζωή σου κατά τέτοιο τρόπο. Καταλαβαίνω τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι ε, τα εθνικά δικαστήρια είναι ο η καλύτερη διέξοδος και ότι μπορεί να μην ε, είναι το, το καλύτερο να πάμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα κάτω αυτή τη στιγμή, αλλά ενδεχομένως ε, να ε, μπορούμε όντω να πούμε ότι είναι πιο αρμόζον να επιληφθεί το τοπικό και περιφερικό επίπεδο, αλλά επειδή είναι ευρωπαϊκό το θέμα, ε, και επειδή πρόκειται για παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλει επιστολή στον ε, Ισπανό ε, ρυθμιστή, ρυθμιστή περιβαλλοντικών θεμάτων, ώστε να λυθεί το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν για τους ανθρώπους τους οποίους δημιουργεί πρόβλημα αυτό το θέμα. Μπορώ να φανταστώ λατομία λίθου στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποθέσεις που τράβηξαν πολλά χρόνια επειδή έμεναν δίπλα σε παρόμοιες εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορώ να καταλάβω την απογοήτευση και την αγανάκτησή τους για το, τη βραδύτητα των διαδικασιών και της επίλυσης των προβλημάτων, να πω ότι ελπίζω η επίλυση να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, συμφωνώντας σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε η Τζουντ. Εγώ λέω να στείλουμε ένα γράμμα στις αρχές της Βαλένθια και του Πέγκο, ε, στις τοπικές αρχές για να εξηγήσουμε την κατάσταση που πραγματικά ε, προκαλεί τεράστιο πρόβλημα ε, στον αναφέροντα βάσει της αναφοράς που λάβαμε και να πούμε ότι η ενωσιακή νομοθεσία, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έτυχε πλήρους σεβασμού και ότι θεωρούμε δεδομένο ότι θα ε, κλείσει αυτό το λατομείο ε, που εξακολουθεί να λειτουργεί παρά το γεγονός ότι υπήρξε απόφαση να κλείσει. Ε, νομίζω επίσης ότι πρέπει να πούμε σε μια επιστολή προς τον αναφέροντα ότι η αναστολή της δραστηριότητας του λατομείου είναι καλύτερο να επιληθεί στα εθνικά δικαστήρια και επίσης να του αναφέρουμε το ζήτημα της αποζημίωσης, το οποίο έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ούτως θα πράξουμε. Α, ναι. Επίσης, ε, βεβαίως, ε, να ε, έρθουμε σε επαφή και με τον εθνικό περιβαλλοντικό ρυθμιστή της Ισπανίας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να τηρήσουμε ενήμερο τον αναφέροντα για τις δικές μας ενέργειες και να του δείξουμε επίσης ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. Ε, αναφορά 533 για το 2012 σε σχέση με ε, την ε, παραγνώριση από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπής ενός ψηφίσματος συγκεκριμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι εδώ ο Χένι Κλάους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ και νομίζω και η Μιλένα Μιχαήλοβα είναι εδώ. Εσείς αποφασίστε πώς ε, θα πάρετε το λόγο και πώς θα διαιρέσετε το χρόνο ομιλία σας. Ευχαριστώ πολύ. Αξιόριμοι ευρωβουλευτές, για το συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας την ε, έντονη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και του αναφέροντος για χρηστή διαχείριση βάσει του άρθρου 298 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 41 της ε, Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για μια ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη αναφορά, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 2 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως απάντησε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 25η 11 του 2010, επομένω η άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι έχει συμμορφωθεί με τι ε, θεσμικέ τη υποχρεώσει. Βεβαίω γνωρίζουμε ότι απατώντας, ε, ανταποκρινόμενοι σε αυτό το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2010, δεν έχει ε, προτείνει όπως είχε άλλωστε ζητήσει το Κοινοβούλιο, έναν κανόνα ε, διαδικαστικό στον τομέα των παραβάσεων παρόλα αυτά. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν παραγνώρισε, δεν το αγνώρισε αυτό το ψήφισμα, γιατί στην απάντησή της το 2011 αποφα... εξήγησε λεπτομερέστατα την τοποθέτησή της σε σχέση με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν βέβαια σε μη νομοθετικό πλαίσιο. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν παραγνωρίσαμε την ε, άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά εξήγησε με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια ε, την τοποθέτησή της επί του συγκεκριμένου αιτήματο και επιτρέψτε μου να επανεπισημάνω τα βασικά σημεία αυτή τη απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απατώντα το Κοινοβούλιο και κατ' επέκταση στον αναφέροντα ότι η διαδικασία παραβάση, την οποία αφορούσε και το αίτημα του Κοινοβουλίου αλλά και η αναφορά είναι τμήμα των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των άρθρων 258 και 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης, όπως άλλωστε έλεγε και το ε, ψήφισμα και η αναφορά. Συνεπώς ε, δεν μπορούν να τροποποιηθούν οι αρμοδιότητες που ήδη οι συνθήκες δίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Εξήγησε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η διαδικασία παραβάση της Ένωσης όταν εξετάζει αρχές όπως ε, τον ανοιχτό χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία έχουν ε, ήδη, είναι, διέπονται ήδη από ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα πριν, όταν εγκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάση του κανονισμού 1049 του 2001 για την πρόσβαση στα έγγραφα και για άλλα ζητήματα αν δεν υπήρχαν τέτοιου είδου μέσα, ε, θα αποτελούσαν τμήμα αυτού του κώδικα, όπω για παράδειγμα υποχρεώσει ε, ε, αμεροληψία, αντικειμενικότητας, ανάγκη αιτιολόγησης θέσεων, όπως επίσης να εξηγεί αν υπάρχει δικαίωμα έφεσης ή της ύπαρξης συγκριτικής αξιολόγησης για κάποιες συγκεκριμένε δράσει, βάση όλων αυτών, η τη υπαρξη συγκριτικη αξιολογηση για καποιε συγκεκριμένε δρασει βασει ολων αυτων η ευρωπαικη επιτροπη έχει τον δικό της τομέα, ε, τον δικό της κώδικα διοικητικής συμπεριφοράς. Να σας υπενθυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2012, μετά, επαναλαμβάνω, μετά την αναφορά και μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση όσον αφορά τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα ε, στην περίπτωση παραβίασης ενωσιακής νομοθεσίας και σε αυτή την ανακοίνωση προστατεύει την θέση του καταγγέλλοντος στην ανεπίσημη φάση μιας ε, επιπαραβάσης διαδικασίας, μεταξύ των οποίων τα μέτρα περιλαμβάνουν ε, μια δωδεκάμενη προθεσμία από την αρχιοθέτηση της καταγγελίας, εντός της οποίας προθεσμίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά γενικό κανόνα πρέπει να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει διαδικασία επιπαραβάση. Η πιθανότητα ε, συνάντησης ε, του καταγγέλλοντος με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης υπάρχει για να παρουσιάσει την επιχειρηματολογία του και επίσης πρέπει να δοθεί και πρώτερη ειδοποίηση αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να κλείσει μια υπόθεση δίνοντας την ευκαιρία στον καταγγέλλοντα να παραθέσει νέα επιχειρήματα εντός τεσσάρων εβδομάδων. Λαμβανομένων λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων Απαντώντας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2011, συμπέρανε ότι δεν χρειαζόταν ένα νέο νομοθέτημα για, ε, μια, ε, για, ένα, σύνολο κανόνων διαδικασία στην περίπτωση παράβασης. Δύο πάρα πολλοί γενναίοι συνάδελφοι εξακολουθούν να παρίστανται Θέλει κανείς να πάρει το λόγο ή να προτείνει τίποτα για το πώς να προχωρήσουμε. Αν όχι, να προτείνω εγώ κάτι. Νομίζω ότι έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε λέω αυτή την ανακοίνωση που αφορά την ε, ενημέρωση ε, της ε, των της διαδικασίας επί του 2012, να την αποστείλουμε στον αναφέροντα ενημερωτικά και μετά να κλείσουμε την αναφορά. Νομίζω ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Τζούντ, έχει το λόγο. Συμφωνώ. Συμφωνώ με την πρότασή σας. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πάρα πολύ καλό που υπάρχουν πολίτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διαβάζουν τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα υπερασπίζονται και ενεργά ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήταν πάρα πολύ καλό αν όλα τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου ε, είχαν τόσο καλά στοιχεία ε, από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπής που να, να, να ενημερώνονται δηλαδή τόσο πολύ, να τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνουν τα ψηφίσματα αυτά και νομίζω ότι θα έπρεπε να το πούμε και αυτό στον αναφέροντα. Κυρία Πιτέρα. Άλλο ο Πιτέλα, άλλο είναι ο Πιτέλα, αλλά έχει προχωρήσει και η ώρα. Η κυρία Πιτέρα. Λοιπόν, είμαι θετική όσον αφορά αυτή την τοποθέτηση. Είναι η καλύτερη λύση και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμο να διαβάζει αυτά τα έγγραφα. Το ήθελα να πω και ευχαριστώ. Και αν τα διαβάζουν τα έγγραφα πρέπει να είναι και φιλικά προς το χρήστη. Το θεωρώ και αυτό σαν ένα σημείο ε, έμπνευση που βγαίνει από τις συνεδριάσεις Δηλαδή στο μέλλον να είναι φιλικές προς το χρήστη οι ανακοινώσεις, ούτως ώστε μαζί με ένα συνοδευτικό γράμμα ε, με τα χαράς να μπορούμε να, το, να στέλνουμε τις επιστολές, να επιβάζουμε και στους πολίτες Ευρώπης. Δοθήσεις της αρίστης συνεργασίας μας, σίγουρα αυτό θα ισχύσει. Έτσι δεν περαιτέρω στο μέλλον. Ευχαριστώ όλους σας. Φτάσαμε στο τέλος. Έχετε σχεδόν 50 λεπτά για να χαλαρώσετε από ότι την κανονική λήξη. Τελειώσαν 50 λεπτά νωρίτερα με άλλα λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και η τελευταία συνεδρίαση πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Σας ευχαριστώ για αυτό το εξάμεινο. Σας ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε. Συνδρομή σας στην Επιτροπή. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχιζόμενη πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του προσωπικού, του συμβούλου πολιτική, του βοηθού και σίγουρα θα συναντηθούμε στου διαδρόμου. Αν όχι, επισήμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμό σε καινούριου χρόνου.